Σήμερα έχουμε γεμάτο αλλά ενδιαφέρον πρόγραμμα. Έχουμε συζητήσεις για το θέμα της έρευνας. Και πριν περάσουμε στα συγκεκριμένα έργα, έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα στον τομέα της έρευνας που μπορούν να μας κάνουν λίγο πιο ενημερωμένους για τις εξελίξεις. Έχουμε το σημείο 9 πρώτα απ' όλα, το Ευρωπαϊκό του Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Θέλουμε να συζητήσουμε βεβαίως με τον Διευθυντή ε, του Ευρωπαϊκού του Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την κατάσταση και καλωσορίζω τον κύριο Ρόναλτ Τεμπρούν και τον καθηγητή Μάριο Ρίτερ, Βίλεμ Γιόνκο, ξέχασα κάποιον, και τον κύριο Διέγκο Παβία. Συμφωνήσαμε πως καθένας από τους τέσσερις θα έχει γύρω στα 10 λεπτά για να κάνει μία παρουσίαση θα στριμωχτούμε λίγο, αλλά μπορεί να μας βοηθήσει κιόλας και μετά θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε και ερωτήσεις. Αν α, συμφωνείτε, θα προχωρήσουμε έτσι, οπότε να δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Ρόναλντ Ντεμπρίν. Σας καλωσορίζω όλους. Αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία ήταν στην αρχή επίμαχα, αλλά βεβαίως μετά γίνανε πιο συνενετικά. Έχετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να σας μιλήσω για το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το EIT, και να σας μιλήσω και για τα εταιρικά μας σχέδια. Let's see if the technology doesn't die on us. να μην μας εγκαταλείψει η τεχνολογία. Ωραία. Βλέπετε γιατί χρειαζόμαστε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Είμαστε πολύ καλοί στην έρευνα ως Ευρωπαίοι, αλλά δεν προσφέρουμε πολύ καλά ε, αποτελέσματα στην αγορά. Άρα ε, υπάρχει επιβράδυνση στη ε, στην καινοτομία σε σχέση με, τους, ε, με τη ΣΥΠΑ. Το Ινστιτούτο δεν είναι μηχανισμός χρηματοδότησης. Είναι η πρώτη πρωτοβουλία στην Ευρώπη όπου συμμετέχουν και τα τρία μέρη του τριγώνου της γνώσης. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, για πρόκειται τις επιχειρήσεις, τα κέντρα έρευνας και τον ε, τομέα της εκπαίδευσης, της υψηλότερης εκπαίδευσης και σε σχέση με τη, τα επιχειρηματικά σχέδια χρειαζόμαστε περισσότερο input, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι να αποτελέσουν και την επόμενη γενεά επιχειρηματιών. Σας μίλησα για τα KICS, για τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Τα KICS έχουν συγκεκριμένα στοιχεία, είναι αυτόνομα, ε, αυτόνομα από νομικής πλευράς αυτές οι κοινότητες υπό την ηγεσία ενός διευθύνοντος σύμβουλου. Έχουμε τρεις ε, τομείς που μας απασχολούν. Το θέμα του κλίματος, τον τομέα των ε, τεχνολογιών, πληροφοριών και επικοινωνίας και την, ε, τον τομέα της ενέργειας. Τα ΚΙΚΣ βασίζονται σε σημεία καινοτομίας. Κάθε ΚΙΚ έχει πέντε με έξι hot spots και τα βλέπετε αυτά τα σημεία στη χαρτογράφηση. Βλέπετε εξ αρχής ότι υπάρχει ε, γεωγραφική κάλυψη, αλλά υπάρχουν και πολλά κενά στην κάλυψη. Τι έχουμε κάνει μέχρι τούδε. Θεωρούμε ότι έχοντας να κάνουμε με μία αδυσόπιτη αλυσίδα ε, λάθους και εκπαίδευσης, φτάσαμε στη συγκρότηση της, ε, δική μας, της δικής μας υποδομής με ένα διοικητικό συμβούλιο και με τα ΚΙΚ και τους διευθύνοντες συμβούλους έχουμε τρεις εταιρικές σχέσεις μέσα στα πλαίσια ενός επταετούς προγράμματος. Αυτές οι συμφωνίες πλαίσιο, εταιρικές συμφωνίες πλαίσιο αποτελούν μία μακροχρόνια δέσμευση έτσι ώστε να δημιουργήσουμε νέα καινοτόμα σχήματα μέσα στα πλαίσια των ΚΙΚΣ. Πέρα από αυτό, αρχίσαμε μαζί με τα ΚΙΚΣ να συζητάμε για επιχειρηματικά σχέδια ως προς την εκπαίδευση και την δημιουργία επιχειρήσεων. Ως προς την εκπαίδευση, θα ήθελα να σας πω ότι δύο εβδομάδες πριν είχαμε μία, μία ομάδα ε, φοιτητών από τη Βουδαπέστη και τους είπαμε πόσοι σπουδάζετε για να αποκτήσετε μια θέση εργασίας γέλασαν και μας υπόθηκε ότι φοιτούν για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, κάτι το οποίο δεν είχε σκεφτεί ποτέ κανείς μέχρι τώρα. Αν δείτε τον τομέα λοιπόν της δημιουργίας, ε, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με το MIT είχαν έναν από τους διευθυντές στη Βουδαπέστη και το MIT έρχεται στην Ευρώπη για να δημιουργήσει επιχειρήσεις. Αυτό το πνεύμα πρέπει να μας διέπει και εμάς. Μαθαίνουμε από την πράξη. Λοιπόν, μιλάμε για μία επταετή διεργασία με τα ΚΙΚΣ και δημιουργούμε και ένα στρατηγικό outlook για το 2014 και μετά που συμπίπτει με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Άρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του EIT προσπαθεί να φτάσει σε μια ατζέντα στρατηγικής καινοτομίας, κάτι το οποίο θα σας επεξηγήσω. Πρόκειται για ένα έγγραφο που μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με βάση μια ανοιχτή διαβούλευση και την αποτίμηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας θα προβάλλει την ατζέντα καινοτομία που θα λάβετε εσείς μέχρι το τέλος του έτους από, το από κοινού το Συμβούλιο ένα από τα βασικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας, του EIT, είναι η απλούστευση. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία learning by doing, δηλαδή εκμάθηση μέσα από την πρακτική. Έχουμε κάνει ορισμένα μικρά βήματα στην τροποποίηση των ε, δημοσιονομικών κανόνων, έτσι ώστε να έχουμε ορισμένα καταποκοπήν ποσά τα οποία να διατίθενται στον κεντρικό κορμό των εργασιών μας. Άρα η απλούστευση είναι ένα βασικό στοιχείο. Εμείς Είμαστε ένα αυτόνομο Ινστιτούτο, το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη, χρησιμοποιώντας τα μέσα που προέρχονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό και από τις επιδοτήσεις του. Ε, έχουμε λάβει και ορισμένες εξαιρέσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε επιπρόσθετη χρήση αυτών των επιδοτήσεων με μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά μέσα σε αυτό το κουτί και αυτό θέλει να σας δείξει αυτή η διαφάνεια, είναι ότι υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών. Καθίστατε όμως σαφές ότι αυτά τα πλαίσια δεν οδηγούν σε απλούστευση κανόνων, αυτή η διακριτική ευχέρεια δηλαδή. Άρα συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε κάτι άλλο με βάση το ε, ρόλο μας στα πλαίσια της στρατηγικής ατζέντα και καινοτομίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας υπό την παρούσα μορφή του και μέσα στα πλαίσια της μοναδικότητάς του παρέχει επιδοτήσεις και υποτροφίες και βοηθούμε με κεφάλαιο για πνευματική εργασία να συνεργαστούμε με τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας, τα KICS. Αυτή η ε, ατζέντα στρατηγικής καινοτομίας, όπως την αποκαλούμε, έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή, να λάβουμε υπόψη επενδύσεις ε, οι οποίες να βασίζονται σε επιχειρηματικά σχέδια ως προς ε, χρήματα τα οποία στη συνέχεια μας επιστρέφονται με άλλη μορφή γιατί έχουμε καλύτερα εκπαιδεμένους ανθρώπους και περισσότερες επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο φιλοδοξεί να προωθήσει ένα νέο κύκλο επενδύσεων από το 2014 και μετά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το ρόλο του επενδυτή και με βάση τις επιδοτήσεις και υποτροφίες, αν δείτε τη λογική που μας διέπει εκτός κουτιού, υπάρχει μία πρόταση για έναν χρηματοοικονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επέτρεπε και άλλα είδη χρηματοδότησης, όχι μόνο δηλαδή ε, επενδύσεις, equities ή ε, υποτροφίες επιδοτήσεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του EIT έχει δημιουργήσει το Ίδρυμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας μέσα στα πλαίσια των ΚΙΚΣ, των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, με χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του EITF συνήλθε δύο ή τρεις φορές. Προσπαθούμε λοιπόν να προσδώσουμε, να δώσουμε μια προστιθέμενη αξία στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Μίλησα για την ατζέντα στρατηγικής καινοτομίας. Εδώ έχετε ένα δελτίο που μπορεί να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Ένα πιο εμπεριστατωμένο έγγραφο θα υποβληθεί στις 30 Ιουνίου. Ένας από τους ε, τομείς συζήτησης, ένα από τα θέματα συζήτησης είναι πού θα πρέπει να επενδύσει κανείς. Από το 2014 υπάρχουν ε, διάφορες οδοί που διανοίγονται και που μπορούμε να επιλέξουμε. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την εξής θέση. Πρόθεση είναι να συνεχίσουμε με τις επενδύσεις στα τρία προϋπάρχοντα ΚΙΚΣ, στις τρεις προϋπάρχουσες κοινότητες γνώσης και κοινοτομίας δηλαδή και προσπαθήσαμε να ε, ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Μπορώ να σας μιλήσω για ορισμένους τομείς που πρότεινε το Διοικητικό Συμβούλιο και που συζήτησε με τους εμπλεκόμενους φορείς ε, για την ανθρώπινη ζωή και η υγεία, ε, συνεχή εκπαίδευση, κινητικότητα, ευφυής πόλης, ασφάλεια και υγεία, υγιεινή και ούτω καθεξής. Γνωρίζουμε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν και γι' αυτό χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές. Για να επιλέξουμε λοιπόν τις κοινότητες γνώσης θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούν να κινηθούν πέρα από τον προγραμματισμό έτσι ώστε να εμπλέξουν φορείς και από τα τρία μέρη του τριγώνου δημιουργώντας επιχειρηματικότητα, εκπαίδευση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις. Δηλαδή μας ενδιαφέρει μία εκκίνηση του όλου πλαισίου. Αυτό βεβαίως ε, μας οδηγεί στο να δούμε τη σχέση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας με βάση όλες τις άλλες ε, πρωτοβουλίες. Πιστεύουμε ότι θα ήταν ε, σκόπιμο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο τεχνολογίας να το λάβουμε υπόψη και να το εντάξουμε μέσα στα πλαίσια της έρευνας και καινοτομίας του κοινού στρατηγίου πλαισίου έρευνας και καινοτομίας για να φτάσουμε στην επόμενη γενεά επιχειρηματιών. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα σαφές είναι ότι επειδή υπάρχουν κοινά κέντρα θα πρέπει να αναζητήσουμε συνέργειες με τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για να έχουμε διάδοση πληροφοριών και ούτω καθεξής. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι και το τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να ε, περάσετε στους ε, ενδιαφερόμενους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπούμε που δεν μπορείτε να μιλήσετε περισσότερο. Περνάμε στον επόμενο μιλητή. Η κυρία καθηγήτρια. Um, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε, εμένα και τους συναδέλφους μου, για να μιλήσουμε ενώπιόν σας η καινοτομία για την ευημερία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα είναι ένας από τους βασικούς στόχους ε, των κέντρων καινοτομίας ε, και γνώσεων. Έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για να καλύψουμε μια ένα ευρύτατο πεδίο και χωρίς να βλέπετε τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου θα ε, βλέπετε ήδη μια μεγάλη επικοινομορφία ανάλογα με τις γεωγραφικές, πολιτικές, κοινωνικές διαφορές. Ε, προσπαθήσαμε να καλύψουμε ολόκληρο το πεδίο έχοντας ε, ε, μεγάλη ποικιλία στα μέλη μας. Συγγνώμη, έχω να σας πω ότι έχω υπογράψει πάρα πολλά χαρτιά σήμερα γιατί έχουμε πολύ άριθμα μέλη. Areas. Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς που μας απασχολούν πρώτον η ανάπτυξη πόλεων χαμηλού άνθρακα και η ε, προσπαθούμε να μειώσουμε κατά 70% την εκπομπή του διοξιδίου στην ατμόσφαιρα. Δεύτερος τομέας, ε, η διαχείριση των υδάτινων πόρων, ε, ανάλογα με το αν υπάρχει πλεόνασμα ή έλλειμμα υδάτινων πόρων. Τέταρτη περιοχή, συστήματα παραγωγής ε, μηδενικού άνθρακα ή ελαχίστου άνθρακα ή και αρνητικού, δηλαδή σε ορισμένους τομείς για διάφορα υλικά κατασκευής, όπως το τσιμέντο παραδείγματο χάρη. Ε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν είναι να εκπληρώσουμε τους στόχους μέχρι το 2050. Τέλος, για τη μέτρηση των κλιματικών αλλαγών και των βασικών αιτιών θα πρέπει να έχουμε ε, ενιαία ανάλυση όλων των μετρήσεων, ε, αλλιώς δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης. Βλέπετε το τρίγωνο της γνώσης εδώ πέρα, η έρευνα, οι επιχειρήσεις ε, και η παιδεία και στο κέντρο η καινοτομία. Έχουμε τέσσερις πυλώνες, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα συγκεκριμένα, την παιδεία και τη διερεύνηση νέων λύσεων. Ε, δημιουργούμε νέες συνεργασίες στα πλαίσια του Climate Kick και νέους σχηματισμούς στην αλυσίδα της ε, προστιθέμενης αξίας. και η κοινότητα μας και ο χώρος εργασίας μας χαρακτηρίζεται από το επιχειρηματικό πνεύμα και από την ποικιλομορφία στους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα δημιουργώντας νέους κόμβους ε, επιχειρηματικότητας και επίσης προωθούμε την επιμορία με χαμηλή κατανάλωση του άνθρακα όπως σας έλεγα προηγουμένως δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη καινοτομία. Ε, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα αργότερα. Ε, Επίση, ε, για την διαδικασία της ολοκλήρωσης από τις μεγάλες βιομηχανίες, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα, συγκεντρώνονται διάφοροι φορείς σε αυτές τις πλατφόρμες ε, και έχουμε διάφορους χώρους εργασίας ε, για τις ε, συναντήσεις μας όπου συστεγάζονται διάφορες υπηρεσίες στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ράνστορ και στη Ζηρίχη έχουμε τέτοια κέντρα συστέγαση. Τώρα, αυτή είναι η εκδοχή ΚΙΚ του πρώτου χάρτη. Έχουμε πέντε τέτοια ε, κέντρα συστέγασης. Τα βλέπετε με το πράσινο, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, επιπροσθέτως βλέπετε τις κίτρινες κουκιδίτσες ε, που εκπροσωπούν ε, τα περιφερειακά κέντρα καινοτομία που έχουμε. Είναι ομάδες μικρών βιομηχανιών, αυτοδιοικητικών αρχών και ερευνητικών ιδρυμάτων που μας βοηθούν να εισχωρήσουμε και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, σε Μίλια στην Ουγγαρία, τέλος πάντων σε διάφορα μέρη, στην Πολωνία και στα Ανατολικά Midlands, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Our partners. We have... Οι εταίροι μας, 20 είναι βασικοί. 50% περίπου από ε, τον επιχειρηματικό κόσμο και 50% από τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια. Έχουμε εταιρείε όπως η EDF, η Bayer, DSM, το αεροδρόμιο του Skiphol, GDF Suez και τα λοιπά και μεγάλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Imperial College, ε, TU Delft και τα λοιπά όπως βλέπετε στη διαφάνεια. Θα σας δείξω τώρα τις ε, έξι περιοχές που ε, δημιούργησαν αυτά τα κέντρα, αλλά μην ξεχνάτε ότι πάντοτε υπάρχουν πολλοί άριθμοι εταίροι. Ε, έχουμε επίσης 65 συνδεδεμένα μέλη και οι 32 συνδέονται με τα πέντε κέντρα συστέγασης και οι 35 συνδέονται με τα περιφερειακά με τις περιφερειακές κοινότητες, τα περιφερειακά κέντρα καινοτομία. Ε, πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αυτοδιοικητικές αρχές και μεγαλύτερα θεσμικά όργανα. Για να προσθέσω λίγο κάποιες λεπτομέρειες ε, για τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας. Ε, εκατοντάδες ενότητες βρίσκονται ε, παντού στην Ευρώπη. Έχουν δίκη, τους Διευθυντική Επιτροπή που λειτουργεί ως Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου και καθοδηγεί ε, τις δραστηριότητες ε, του Κέντρου Καινοτομίας. Ε, είναι ένα πολύτιμο πείραμα για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε την καινοτομία και έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Επίσης, μας τροφοδοτούν με πληροφορίες σχετικά με το τι χρειαζόμαστε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και είναι και μοναδική ευκαιρία για ε, φόρου ζωή κατάρτιση. Παραδείγματο χάρη, έχουμε ένα σχετικό πρόγραμμα που έτρεξε πρώτη φορά πέρσι και είχαμε 59 ιδιώτε ε, που έρχονται κυρίω από ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει και ήθελαν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία, ούτω ώστε να προωθήσουν περαιτέρω στον επιχειρηματικό κόσμο την επιχείρησή του για μια σε περίοδο 12 μηνών θα ε, πάνε σε τρία διαφορετικά κέντρα που θα επιλέξουν. Παραδείγματο χάρη, ή σε με μεγάλε επιχειρήσει, αν προέρχονται από μικρομεσαίε επιχειρήσει, ή μπορεί να πάνε σε κάποιο ερευνητικό ίδρυμα για να δουν τι τελευταίε έρευνε που γίνονται, ή, εν πάση περιπτώσει, να πάνε σε κάποιο ε, πολιτικό όργανο για να δουν πώ εφαρμόζεται η νομοθεσία και στις συνέχεια ε, γίνεται η ανταλλαγή απόψεων στις συναντήσεις. Ε, βλέπετε είναι σαν ομόκεντρη κύκλοι και έτσι διαχέουμε τα ευχάριστα νέα και τις ε, πληροφορίες για όλους όσους συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Well. Πώς οργανωνόμαστε λοιπόν για να δούμε. Η έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και την Κοινότητα. Για να τα δούμε ε, με μεγαλύτερε λεπτομέρειε. Σα μίλησα για του εταίρου, για τα συνδεδεμένα μέλη. Όλοι υπομίζονται την ευθύνη για τα χρήματα ε, που λαμβάνουν, ε, αλλά η βασική μα εταίροι αναλαμβάνουν την ευθύνη και για τι νομικέ οντότητε. Τα συνδεδεμένα μέλη εκπροσωπούνται, ενώ τα βασικά μέλη είναι πλήρη μέλη. Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο ε, απαρτίζεται από 11 μέλη, δύο από κάθε κέντρο συστέγασης ε, και από τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας. Εκπροσωπούνται έτσι οι περιοχές και όχι τα θεσμικά όργανα σε επίπεδο ΚΙΚ. Μία φορά το χρόνο συναντιόμαστε όλα τα μέλη δηλαδή, της κοινότητας ΚΙΚ και διοργανώνουμε το φεστιβάλ που τώρα για φέτος θα γίνει στη Βουδαπέστη, τέλη Σεπτεμβρίου. Ε, για το επιχειρηματικό μας ε, σχέδιο για την εφαρμογή του χρησιμοποιούμε τους τέσσερις πυλώνες ε, και έχουμε και το οικολογικό σύστημα όπου αναπτύσσουμε τη δράση κάθε πυλώνα. Είναι συνεταιρική διαχείριση. εγώ είμαι εκτελεστική σύμβουλος και έχω και διευθυντή των επιχειρήσεων που με επικουρεί στα καθήκοντά μου. Τι κάνουμε στο ΚΙΚ. Οι ε, εταίροι από όλου τους διαφορετικούς ε, κλάδους ε, συναντιούνται και εστιάζουν την προσοχή τους κατά προτεραιότητα σε αυτά τα τέσσερα βασικά θέματα που ανέφερα στην αρχή και μετά κατανοούμε τις δραστηριότητες σαν πυλώνα, καινοτομία είπαμε, διαρευνητικός πυλώνας, παιδεία και έρευνα και τέλος θα ήθελα να σας περάσω τρία μηνύματα από πέρσι Φυσικά ε, έπρεπε να αναδιοργανώσουμε τη δομή μας, να οργανώσουμε αυτά τα κέντρα συστέγασης και χάσαμε λίγο χρόνο, αλλά παρόλα αυτά έχουμε συνεργαστεί με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολύτιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε ε, τη στρατηγική μας. Σας μίλησα για τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας που ιδρύθηκαν πέρσι και τέλος ε, για του, όσους κάνουν διδακτορικό έχουμε οργανώσει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι και πριν αρχίσουν περνάνε έξι μήνες επί το όπου δηλαδή πηγαίνουν σε τρία από τα κέντρα συστέγασης και γίνονται διαλέξεις όπου τους παρουσιάζονται τα βασικά θέματα, αλλά όχι μόνο, συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και αναλύουν τις πληροφορίες, προτείνουν επιχειρηματικά ε, προγράμματα. Ε, και στι ομάδες εργασία υπάρχει και ανταγωνισμό μετά τι έξι εβδομάδες ε, ε, δύο από αυτού που κέρδισαν βραβείο πήραν και επιχορήγηση για δύο επιχειρήσεις μία επιχείρηση κομποστοποίηση παραδείγματο χάρη στην Ουγγάντα και μία άλλη στην Ελβετία και 59 από τους εταίρους μας έχουν συμμετάσχει σε ε, πρακτική και ελπίζουμε στο μέλλον να συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα και να πολλαπλασιαστούν τα μέλη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω μέσα τον λόγο στον κύριο Διέγκο Πάβια χωρίς να μακρηγορήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας ε, κύριες ε, και κύριοι. Εγώ θα μιλήσω για την ΚΙΚ στην ενέργεια. Ποια είναι η αποστολή μας. Είναι να αποτελέσουμε ένα κινητήρα καινοτομία για η φόρο ενέργεια. Και εδώ μιλάμε για έξι δραστηριότητες. Δηλαδή βασιζόμαστε στον καθαρό ε, άνθρακα στα εφή δίκτυα, στις εφή πόλεις, στα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την χρήση των ε, ανανεώσιμων μαζί με την πυρηνική ενέργεια, τη σύγκληση των δύο, καθώς και τα χημικά καύσιμα. Στην ενέργεια κάνουμε ό,τι άλλο θέλετε εκτός από την καύση και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε ως προς τις ανάγκες μας. Μιλάμε για 700 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψουμε τους έξι αυτούς τομείς. Γι' αυτό επειδή είμαστε μια εταιρεία με μετόχους, 29 μετόχους, ε, έχουμε προωθήσει ένα επταετές πρόγραμμα. Και μόνο τα τέσσερα πρώτα χρόνια αφορούν μία επένδυση της τάξης των 700 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2011 και 2015. Μιλάμε λοιπόν για τη μόχλευση 700 εκατομμυρίων ευρώ που θα πρέπει να προέρχονται από τους επενδυτές. Οι δραστηριότητες μας σχετίζονται με τους τρεις στόχους. Ή θα μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, ή θα αυξήσουμε την ε, ασφάλεια ή θα μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου, ε, ε, αερίων του θερμοκηπίου, με συγχωρείτε. Είτε έναν από τους τρεις τομείς, είτε δύο, είτε και τους τρεις. Εάν μπορέσουμε να μειώσουμε κατά 1% το κόστος της ενέργειας σήμερα την Ευρώπη, θα είχε επίπτωση 20 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμησης. Αυτά τα 20 εκατομμύρια λοιπόν δημιουργούν σε επιπρόσθετη ανταγωνιστικότητα για τη βιομηχανία ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θύλακας ευημερία. Δηλαδή με μείωση κόστους ενέργειας κατά 1% θα είχαμε 20 δισεκατομμύρια ευρώ εξοικονόμησης και μιλάμε για τις τρεις βασικές δραστηριότητες, την εκπαίδευση, τα τεχνολογικά ε, σχέδια που να βρίσκονται πολύ κοντά στην αγορά και να δημιουργήσουμε επιχειρηματίες με βάση τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία, αν θα μπορούσα να τα πω να τα κατονομάσω έτσι, της ε, τεχνολογίας. Βασιζόμαστε στο ταλέντο στους ανθρώπους και όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι δόκτορες, οι μηχανικοί θα κατέχουν αυτή τη τεχνογνωσία και θα μπορούσαν και οι ίδιοι να προωθήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ξεκινάμε από τους φοιτητές αλλά και με την διαβίου μάθηση δηλαδή τους επιχειρηματίες που βρίσκονται στο μέσον της σταδιοδρομίας τους. Ποιος θέλει να αγοράσει αυτές τις υπηρεσίες από τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να χρησιμοποιήσουμε τους προϋπάρχοντες μηχανισμούς για να υπογραμμίσουμε αυτά τα μηνύματα. Άρα, τι κάνουμε, χρησιμοποιούμε την ενέργεια με βάση τα κίξ. Τις ε, κοινότητες γνώσης και στόχος είναι να έχουμε 160 φοιτητές το Σεπτέμβριο. Έχουμε 650 υποψηφίους για αυτά τα νέα project. Άρα οι φοιτητές που θέλουν να αδράξουν αυτά τα μάστερ μπορούν να το κάνουν. Οι τομεί αυτοί είναι διαφορετικοί διότι αφορούν όχι μόνο την βασική και παραδοσιακή εκπαίδευση αλλά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό τομέα. Και μιλάμε βεβαίως για συνεργασία με κοινοπραξίες. Επίσης, το 55% αφορά σχέδια τεχνολογίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μία ευρωπαϊκή προσπάθεια. Η κάθε οριζόντια γραμμή, δηλαδή 31 ε, ε, γραμμές για το 2011, θα αφορούν τις καλύτερες επιδόσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι η δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Ήδη από το Σεπτέμβριο Μέχρι τώρα τρία ε, projects δεν έγιναν αποδεκτά διότι δεν ήταν στο ύψος των προσδοκιών μας. Δηλαδή να βασίζονται σε στοιχεία αριστείας. Τρίτον, επιχειρηματικότητα. Χρησιμοποιούμε πολλούς ε, επιχειρηματίες ή ε, ανθρώπους που κατέχουν τεχνογνωσία, επιστήμονες, έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν σχέδια και να τους βρούμε και τον πρώτο τους πελάτη. Και όλες μας οι υπηρεσίες ε, είναι, ε, παρέχονται δωρεάν μέχρι να συσταθεί η επιχείρηση. Αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ότι το 8% αφορά τον ε, δικό μας προϋπολογισμό. Και έχουμε ξεκινήσει με ένα πανεπιστήμιο ε, για ντοκτορά. Δύο από αυτούς τους φοιτητές έχουν ξεκινήσει με νεοσύστατες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τον κύκλο της ε, τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της δημιουργίας επιχειρήσεων με βάση την εκπαίδευση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, είναι η επιχείρηση να λειτουργεί καλώς και οι επενδυτές που δεσμεύτηκαν για 7 χρόνια να δουν συγκεκριμένη απόδοση. Βλέπουμε δηλαδή ε, ε, την έρευνα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση. Βλέπετε λοιπόν πόσες επιχειρήσεις συμμετέχουν. 44 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα όχι μόνο ε, στα ε, πλαίσια των, ε, των αλλά και στα πλαίσια των μικρομεσαίων. Τι γίνεται σε σχέση με τα KPI. Αν δεν ανταποκριθούμε στα KPI, τότε τι θα γίνει. Θα με απολύσουν εμένα προσωπικά αν δεν ανταποκριθώ στα KPI. Άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κερδοφορία, προς τα εκεί προσανατολιζόμαστε. Και θα πρέπει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προδιαγραφές, αυτού δηλαδή του scoreboard. Να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και να προβάλλουμε ε, κερδοφορία μέχρι 28 KPIs. δεν βρισκόμαστε στην έρημο. Θα πρέπει να υπάρξει διάδραση με άλλους φορείς, γιατί όλοι βρισκόμαστε στον ίδιο τόπο δράσης. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με τα κοινά κέντρα ερευνών, με βάση τις θεματικές που προβάλλονται δηλαδή προσωμείωση για μελλοντικά σενάρια έτσι ώστε να δώσουμε επιστημονικά και πραγματιστικά στοιχεία σε αυτούς που ε, καταρτίζουν την πολιτική. Τα ΚΙΚ αφορούν ένα από τα θεματικά μας, ε, ε, τους θεματικούς μας κύκλους σε συνεργασία με τα κοινά κέντρα ερευνών. Δεν έχουμε ακόμα ορίσει όλα τα σχέδια με τις άλλες γενικές διευθύνσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τελευταίος ο καθηγητής Βίλεμ Γιόνκα, ο οποίος έχει τελευταίως την ευκαιρία να μιλήσει. Terwijl de presentatie wordt opgebracht, allereerst eh, meneer de voorzitter, eh, dank voor uw uitnodiging. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, πρόσκλησή σας. Θα συνεχίσω στα αγγλικά για να βγάλετε και τα ακουστικά σας, μη φοβάστε. Να σας πω κάτι για το πώς έχουν τα πράγματα στα εργαστήρια πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Πρώτα απ' όλα το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό Πολυτεχνείο θα λέγαμε υπάρχει, η κεντρική διοίκηση υπάρχει και πριν από τρία χρόνια θα έλεγα δεν σκεφτόμασταν πως αυτό θα συνέβαινε σήμερα. Και όμως είναι μια πραγματικότητα και αυτό είναι φοβερό επίτευγμα. Υπάρχουμε, λειτουργούμε, αλλά μπορείτε επίσης να δείτε πως είμαστε και νέοι. Από τον Οκτώβριο πέρσι ε, έχουμε νομική προσωπικότητα και υπογράψαμε μια σύμβαση πλαίσιο μόλις το Δεκέμβρη και έχουμε Μάιο Μιλάμε για το, πραγματικό, πρώτο πραγματικό, το πρώτο έτος πραγματικής λειτουργίας. Ένα από αυτό το οποίο, τα πράγματα τα οποία δεν είχαν συνειδητοποιήσει οι άνθρωποι είναι το πώς αλλάζουν οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ε, της ζωής σας. Δεν ξέρω αν ε, ε, ξέρετε βεβαίως πώς, δεν ξέρω αν ξέρετε πώς χρήστες έχει ε, το Google σήμερα πριν από 12 χρόνια δεν υπήρχε και δεν ξέρω πόσα παράπονα έχετε για τα τηλέφωνά σας, τα smartphones και ειδικά για τις μπαταρίες τους, αλλά πριν από λίγα χρόνια επίσης δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω επίσης ε, πόσο συχνά χτυπάτε με τα μάξι σας κάπου, γιατί πλέον έχει το, τους αισθητήρε, αλλά εσείς τους αγνοείτε, αλλά πριν από 10 χρόνια ούτε αισθητήρε υπήρχαν στα αυτοκίνητα. Οι τεχνολογίες αυτές λοιπόν υπάρχουν παντού και αυξάνονται με ρυθμό αλματώδη. Και αν δείτε την τιμή σε σχέση με την ε, απόδοση, είναι φοβερός αυτός ο λόγος, η αναλογία. Και ένας Ολλανδός συνάλφος μου είπε πως ε, εάν έκανε το ίδιο και αυτοκινητομηχανία, η Mercedes ES 500 σήμερα θα κόστιζε 2 ευρώ και θα είχαμε όλοι από μία. Ε, ίσως να μην ήταν τόσο καλό για την ενέργεια βεβαίως και το περιβάλλον. Η αποστολή μας βεβαίως είναι φυγαμισμένη με αυτή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και το σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να υπάρχει ταλέντο. Επενδύουμε στις νέες γενιές, όχι μόνο στις νέες γενιές. Η εκπαίδευση είναι κάτι το οποίο υπάρχει διαβίου. Και εγώ μπορώ να σα πω προσωπικά πως μαθαίνω πολλά κάθε μέρα από αυτή την προσπάθεια. Εκεί υπάρχουμε, έχουμε τέσσερις έδρες, Ελσίνκι, Στοχόλμη, Εντχόβεν, Βερολίνο, Παρίσι και ε, άλλα γραφεία στο Λονδίνο, Τρέντοφ και Βουδαπέστη. Αυτή είναι η εταίροι μας, βλέπω το ολόκληρο κατάλογο, αλλά εντός του δικού μας ΚΙΚ υπάρχουν οι βασικές βιομηχανίες, SAP, Deutsche Telekom, Philips, Siemens, Nokia, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θεωρούμε πως ένα οικοσύστημα αν θέλετε μπορεί να λειτουργήσει αν υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των μεγάλων και των μικρών έχουμε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για να μας βοηθήσουν ε, να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία θέλουμε και να φροντίσουμε η Ευρώπη να παραμείνει στο προσκήνιο των εξελίξεων αυτών. Έχουμε λοιπόν μια γενική συνέλευση, ένα εκτελεστικό συνέδριο και μια διαχειριστική ομάδα. Λειτουργούμε σαν εταιρεία και βλέπετε τη σύνθεση της ομάδας. Το εκτελεστικό συμβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει ε, έναν άτομο από το πανεπιστημιακό τομέα και έναν άτομο, ένα άτομο από την βιομηχανία. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα τους ε, διευθυντέ και αν έχει βεβαίως κανείς μία εταιρεία χρειάζεται και ένα πρόγραμμα διαχείρισης και αν έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να αφιερώσει τον χρόνο του πρέπει ε, να δώσει κάποιες προτεραιότητες για να γίνεται η δουλειά. Έχουμε λοιπόν εμείς πολύ απλές προτεραιότητες, πρέπει να οργανωθούμε και να αναγνωριστούμε. Εάν το έχουμε καταφέρει αυτό μέχρι το τέλος του έτους, εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Και αυτό προσπαθούμε αυτή τη στιγμή μέσω των καταλητών καινοτομία, μέσω των δράσεών μας που δουλεύουμε σε θεματικούς τομείς, σε κοινωνικά προβλήματα όπως η κινητικότητα, ψηφιακές πόλεις του μέλλοντος, διαχείριση ενέργειας κτλ. Και δεν είμαστε μόνοι που δουλεύουμε σε αυτά, γιατί νομίζω πως ο μισός κόσμος δουλεύει πάνω σε αυτά. Είμαστε μοναδικοί όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσής μας που συνδυάζουμε την εκπαίδευση, την έρευνα και τις επιχειρήσεις σε ένα σώμα. Τα κέντρα αυτά, όπως είπαμε, συστέγασης πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε πέντε τέτοια. Είναι υπαρκτά κτίρια, γιατί ακόμα και στον ψηφιακό κόσμο θεωρούμε πως πρέπει να έρχονται οι άνθρωποι σε επαφή. Έχει μια προσθέμενη αξία αυτό. Καθώς οι επαφές στον ψηφιακό κόσμο δεν είναι τόσο πραγματικές, θα έλεγα. Εδώ πέρα έχουμε το πλαίσιο καινοτομία που μα απασχολεί, μοιάζει πολύπλοκη εικόνα, αλλά είναι απλούστατο. Για να είναι κανεί επιτυχή χρειάζεται ταλαντούχου ανθρώπου, καλέ ιδέε και ε, να μπορέσει να τα φέρει όλα αυτά στην αγορά. Γιατί είναι εύκολο να ανοίξει κανεί ένα μαγαζί, αλλά εάν δεν έχει πελάτε, δεν δουλεύει. Έχουμε μια απλοποιημένη εικόνα εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε ταλέντο, ιδέε και πελάτε, αλλά βεβαίως ο τρόπος παραγωγής των ιδεών είναι ο εξή Πρέπει να φροντίσουμε οι ιδέε να είναι εκμεταλλεύσιμες άμεσα. Και εκεί πέρα πρέπει να βελτιωθούμε στην Ευρώπη. Έχουμε εξαιρετικού ερευνητέ εξαιρετικά συστήματα εκπαίδευσης, αλλά το να γίνει αυτό, να μεταφραστεί σε οικονομική αξία, σε θέσεις εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν θέλουμε να τους δώσουμε ταλέντο στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε δουλειές υψηλής αξίας. Μετράμε λοιπόν τα μετράμε KPI, όπως πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή βασικούς ε, δείκτες απόδοσης. Και εδώ πέρα έχουμε κάποιους δείκτες, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με αυτούς τους δείκτες, γιατί είναι πάντα βράχη πρόθεσμα μέτρα. Παραδείγματος χάρη δείτε την εκπαίδευση. Μετράμε τον αριθμό φοιτητών που εγγράφονται, αριθμό υποψίων διδακτόρων. Αλλά ο πραγματικός δείκτης είναι έχ, βγάζουμε πραγματικά κορυφαία ταλέντα. Ε, αυτό θα το ξέρουμε μετά από 10-15 χρόνια και να δούμε πόσοι από αυτούς τους φοιτητές μας κατέληξαν σε θέσεις κλειδιά στον ευρωπαϊκό αυτό τομέα. Αυτό είναι ο δείκτης που αναζητούμε. Αυτό το μοντέλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για έναν καταλήτη ε, για να λειτουργήσει αν θέλετε ως λιπαντικό στην όλη υπόθεση όπως είπε και ο Διέγκο. έχουμε λοιπόν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο επενδύσεων που χρησιμοποιούμε τα λεφτά αυτά ως καταλητικός το κάνουμε π.χ. στην εκπαίδευση έχουμε ένα επιχειρηματικό ένα σύστημα εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα τα συγχωνεύουμε αυτά τα δύο και βγάζουμε το είδος των φοιτητών που θέμε που δεν ε, βρίσκουν μόνο δουλειέ, αλλά δημιουργούν και δουλειέ. Διπλώματα ευρεσιτεχνία. Πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει το σύστημα πιο φτηνό και πιο απλό, αλλά πρέπει και τα ερευνητικά μα έργα να δημιουργούν πολύ περισσότερη πνευματική ιδιοκτησία. Έχουμε συγκεκριμένου καταλήτε που συνδυάζουμε με τα ερευνητικά έργα για να έχουμε περισσότερες, περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνία από την έρευνα. Γιατί δεν δημιουργούνται εταιρείε μόνο από τι δημοσιεύσει, χρειάζονται διπλώματα ευρεσιτεχνία, δηλαδή προϊόντα. Μεταφορέ τεχνολογίες. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολύ τεχνολογία που κυκλοφορεί, πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και το να συγκεράσουμε αυτά τα δύο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει λοιπόν και εδώ πέρα ένα καταλήτη που συνδυάζει τις τεχνολογίες για να μην καταλήγουν τα πράγματα στο ράφι ή στα σκουπίδια αλλά στην αγορά. Θα πω κάποια πράγματα για τις γραμμές δράσης εδώ πέρα. Έχουμε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, αλλά έχουμε και ένα πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να έχουμε μια συμφωνία ετήσιου σχεδίου. Και αυτό μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, να δημιουργήσουμε το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2012. και είδαμε ποιο είναι το δυναμικό καινοτομία που υπάρχει εδώ πέρα και ποια είναι τα χρήματα που έχουμε δώσει στον τομέα των καταλητών, όπως είπα. Θα περάσω αυτή τη διαφάνεια, απλά να πω πώς ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλες ενέργειες, π.χ. με την ε, ΙΤΕΑ είμαστε τώρα σε μια συνεργασία όπου έχουμε τα χρήματα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εθνική χρηματοδότηση του έργου ΙΤΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες βεβαίως υπάρχει η ιστοσελίδα μας. So, ganz Dank. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ε, ήταν συναρπαστικά όλα αυτά. Και... Θέλω βεβαίω να σας δώσω και την ευκαιρία, να δώσω την ευκαιρία στου συναδέλφους να θέσουν ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα λοιπόν η κυρία Καρβάλιο που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα, για τα επιτεύγματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι διαπιστώνω ότι αυτό το πρόγραμμα που ακολουθώ εξ αρχής, με άλλη ιδιότητα βέβαια, έχει επιτυχία. Είναι καινοτόμο διότι προσεγγίζει με ορθό τρόπο την καινοτομία. Δηλαδή η καινοτομία είναι απόρρια του συνδυασμού ε, της παιδείας, ε, του επιχειρηματικού κόσμου και της έρευνας. Δεύτερον, η ανεξαρτησία, η αυτονομία της, ε, του οργανισμού. Και τρίτον, απλούστευση σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα. Because at the moment we ε, τώρα συζητούμε το κοινό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία και άρα θα μας ενδιαφέρε πολύ να ακούσουμε την άποψή σας. Ε, γνωρίζουμε ότι σημειώσατε επιτυχία για την ολοκλήρωση, τη διαδικασία ολοκλήρωσης, αλλά θα ήθελα να μιλήσετε περισσότερο για την ανεξαρτησία και για τη διαδικασία απλούστευσης. Ποια είναι η εμπειρία σας ε, από αυτήν την ανεξαρτητοποίηση από τη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το πλεονέκτημα διότι οι επιστήμονες λειτουργούν ανεξάρτητα, όμως ε, χάνετε την εμπειρία που θα σας προσέφερε μια δομή όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάρη στην οποία εμπειρία θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε περίπλοκα ε, πράγματα, χρηματοδοτικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη και ούτω καθεξής. Δεύτερον, απλούστευση σε σχέση με το ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7 έχετε κάνει αλλαγές. Σας ικανοποιούν. Γιατί ρωτάω, διότι έμαθα, είπατε ότι υπογράψατε τις συμβάσεις σήμερα το πρωί. Ε, θελήσατε να έχετε μία καινοτόμο και απλή δομή. Ε, το καταφέρατε κατά τη γνώμη σας με τους ε, κανόνες που έχετε θεσπίσει ή τώρα που προσπαθούμε να πλουστεύσουμε όλους τους κανόνες για το επόμενο πρόγραμμα έρευνας θα ήταν καλύτερο ε, να θεσπίσουμε κοινούς κανόνες ε, ως προς τη διαδικασία απλοποίησης. Αυτές τις ε, δύο ερωτήσεις θα εκτιμούσα πολύ να μας απαντούσατε, οποιοδήποτε εκπρόσωπος του ΚΙΚ δηλαδή. Ευχαριστώ. Ο κύριος δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να πάρω εγώ το λόγο, διότι ο κύριος Ρούμπιχ δεν είναι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, διευθύνοντες των τριών ΚΙΚΣ. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί βρίσκεστε στην Επιτροπή μας και θα ήθελα και να σας συγχαρώ. Είναι μεγάλο το κέρδος από την παρουσία σας και μπορούμε να προβούμε σε μια ανταλλαγή απόψεων για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ινστιτούτου. Ξέρω ότι χρειάστηκε να επιλύσετε ε, τα περισσότερα από τα προβλήματα που ανέκυψαν όσο καλύτερα μπορούσατε. Και κάθε φορά συμβαίνει αυτό όταν ε, τίθεται σε εφαρμογή κάτι το καινούριο, όπως ισχύει και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Εμείς έχουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για την ε, υποδομή, τη διάρθρωση του EIT, γιατί είναι κάτι που συζητήθηκε κατά τη σύσταση του Ινστιτούτου. Υπάρχει η έδρα στη Βουδαπέστη και στη συνέχεια έχουμε τα ΚΙΚΣ, τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς λειτουργεί αυτή η διασύνδεση και πώς ε, διέπεται ο συντονισμός, από ποιους ε, αναλαμβάνεται ο συντονισμός αυτών των δραστηριοτήτων. Επίσης, τι δεν λειτουργήσε καλά κατά την άποψή σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αλλάξουμε στις ε, μελλοντικέ προτάσεις ως προς την στρατηγική ατζέντα καινοτομίας μας ε, διαφωτίσατε αρκετά και υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να λάβετε υπόψη την διάσκεψη των εμπλεκομένων φορέων. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και να συσταθούν νέες κοινότητες γιατί για μένα δεν είναι απόλυτα σαφές. Σε σχέση με τις ε, επεξηγήσεις που ε, δόθηκαν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ γιατί φαίνεται ότι επιτελείται ένας από τους στόχους του Ινστιτούτου, δηλαδή να εξευρεθούν πόροι και επενδύσεις από τις επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι μπορέσαμε να επιλύσουμε θέματα ως προς ε, τα startups, τις νεοσυσταθήσεις εταιρείες και επιχειρήσεις και θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορέσατε να φτάσετε σε ανθρώπινους, σε εξέβρεση ανθρωπίνων πόρων όπως θα, θα επιθυμούσατε, διότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, όχι μόνο ως προς την ε, χρηματοδότηση, αλλά και στα ίδια τα προγράμματα των επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ξέρω την άποψη και των δύο πλευρών. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απευθύνομαι στον κύριο Ντεμπρίν. Το θέμα γύρας με υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και στα κράτη-μέλη. Υπάρχει και ένα πιλωτικό έργο και μια, καινοτομία, μια συνεργασία καινοτομίες και σε διάφορες υπηρεσίες στην Κομισιόν ασχολούνται με το θέμα αυτό. Οπότε το ερώτημά μου είναι, κόσμος γυράσκει, η κοινωνία γυράσκει, το θέμα είναι όλο και σημαντικότερο και πώς το βλέπετε για την επόμενη προγραμματική περίοδο να αποκτήσει αυτό το θέμα την ε, χρηματοδότηση που του αξίζει. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ε, e, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Και από όσα ακούσαμε, μας ενδιαφέρει περισσότερο η δομή των χώρων εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Κυρία Ρίτερ, θα μπορούσατε να μας πείτε Εάν εσείς επιλέξατε αυτή την δομή βάσει των ενδιαφερόντων σας, διότι αυτά τα κέντρα βρίσκονται σε ευημερούσες οικονομίες Ελβετία, Φινλανδία, Γερμανία κτλ δεν υπάρχουν σε χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ανατολική, η Ευρώπη, η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Πώς ε, ακριβώς ε, δημιουργούνται οι εταιρικές ε, σχέσεις σε αυτές τις χώρες. Next. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση. Παρεμφέρει από την κυρία Γκρότε. Ε, πώς θα συγχρονιστούν τα κικς με τα EIPs. Έχουμε κικ για το κλίμα, έχουμε κικ για τις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, Τώρα έχουμε τις πρώτες ύλες, ε, εταιρικές για την καινοτομία και την γύρανση θα ιδρυθεί και το σχετικό ΚΙΚ. Η Επίτροπος που ήρθε στην Επιτροπή μας δεν αναφέρθηκε στη δημιουργία ΚΙΚ για την υγιή γύρανση, ούτε ανέφερε, ε, αναφέρθηκε καθόλου στο ΚΙΚ που θα βασίζεται στις βιοτεχνολογίες θα θέλαμε να συντονιστούν, να συγχρονιστούν όλες οι διάσπαρτες προσπάθειες που γίνονται, γιατί φοβούμαστε την επικάλυψη προσπάθειων. Μπορείτε να αναπτύξετε αυτό το θέμα, παρακαλώ. Κύριο Σέλερ. Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και εγώ, όπως και οι συνάδελφοι ήταν ε, πολύ ωραίες οι παρουσιάσεις. Να αναφερθώ και εγώ στο ερώτημα της κυρίας Καρβάγιο. Είναι η γυναίκα και πιο ευγενική, αλλά είπε πως ε, δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε την εμπειρογνωμοσύνη της Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει, εσείς μιλήσατε για το ότι βρίσκεται βρίσκεστε στο πρώτο σας έτος και βεβαίως υπάρχει μεγάλη διάθεση από πλευρά Κοινοβουλίου να σας δώσει δυνατότητα να κάνετε λάθη, αλλά το θέμα είναι πώς έχει η διαδικασία αξιολόγησης αυτά τα 7 χρόνια τα οποία αναφέρατε είναι μεγάλο διάστημα. Ποια διαδικασία αξιολόγηση έχετε θέσει στους εαυτούς σας για να μπορέσετε να μετρήσετε αν θέλετε ε, κάτι σε σχέση με κάποιους ε, στόχους. γιατί πράγματι βεβαίω πρόκειται περί ενός νέου ιδρύματο και το θέμα είναι ποιε διαδικασίες ελέγχου έχετε επιβάλει ίδιοι δεύτερον. Το δεύτερο αναφέρεται στι επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Ποια είναι η στάση των επιχειρήσεων σε σχέση με τα kicks αυτά. Μιλήσατε οι ίδιοι για μετοχές. Ο μέτοχος έχει κάποιες προσδοκίες τι θα λέγατε ε, για το, το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων ως προς αυτό και μετά και εσείς τονίσατε όπως κάνουν όλοι τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά βεβαίως με την πολυπλοκότητα αυτών των ζητημάτων και με με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη φύση τους. το ερώτημα σε ποιο βαθμό ε, έχουν ε, τη δυνατότητα να λάβουν μέρος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, σε ένα τόσο πολύπλοκο πρόγραμμα. Είναι κάτι που το κάνετε έτσι για να δείξετε ότι έχουμε και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή πραγματικά υπάρχει κάποια ουσία εδώ πέρα. Και αυτό το λέω γιατί αφενός υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε επίσης πως σε πάρα πολλά έργα έχουμε κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμβολικά για να γεμίσει η ποσόστοση, αλλά το αποτέλεσμα της συνεισφοράς τους δεν είναι και τόσο σοβαρό. Ευχαριστώ κυρία Τράουτμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα δεν θα μιλήσω εξ ονόματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως συνηθίζω, αλλά θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση και να εκφράσω και μια ευχή. Ε, λυπήθηκα διότι πήγα όχι ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά ως ε, εθνική βουλευτές και κατέθεσα καταγγελία στο Δημεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ε, ε, επιλογής, ε, διότι η δική μας αυτοδιοικητική αρχή, όπως και άλλες, άλλες χώρες, στην Ισπανία παραδείγματος χάρη, συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα που ονομαζόταν e-City, σε ηλεκτρονικές πόλεις. Τέλος πάντων, τελικά δεν εγκρίθηκε το πρόγραμμα, αλλά μέσα στην κριτική επιτροπή έγινε μια επιλογή που όμως δημιούργησε προβλήματα. Θα συνοψίσω γιατί είναι, αυτή είναι η βασική διαφορά. Ε, αναφέρθηκε ότι ήταν ενδεχομένως πρόβλημα η παρουσία της ε, εκπροσώπων της Δημόσιας Αρχής για την επιτυχία του προγράμματος. Ε, δεν, δεν παραθέτω, έτσι θα το συνόψισα. Τέλος πάντων έγινε μια συζήτηση ε, σε μια συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών της Επιτροπής ε, Βιομηχανίας για την ε, ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου και είχε προταθεί από τη συνέλφη και κλείνει το, το σύστημα των ΚΙΚΣ και πραγματικά ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα αυτό. Όμως θα ήθελα από πλευρά του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας ε, ένα μήνυμα. Δεν θεωρώ ούτε καλό ούτε λογικό ένα θεσμικό όργανο, ένας οργανισμός που ιδρύεται και κανονικά θα έπρεπε να εκπληρώνει το στόχο του, δηλαδή ε, να μεριμνά ώστε οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές ε, που ε, υποστηρίζουν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και τη δεσμευσή του στην καινοτομία. Όταν λοιπόν δημιουργούν ένα δίκτυο αυτές οι αρχές γύρω από επιχειρήσεις, γύρω από έναν μεγάλο ερευνητικό οργανισμό θα ήθελα να καταλάβω γιατί θεωρήθηκε ε, αυτός ε, τροτό σημείο του προγράμματος. Ο διαμεσολαβητής ε, της Ένωσης ακόμη δεν έχει απαντήσει και θα ε, ήθελα για να επικρατήσει η διαφάνεια να το αναφέρω στη σημερινή μας συνεδρίαση διότι θεωρώ ότι όταν ξεκινάει ένας οργανισμός, όταν είναι νεόκοπος πρέπει να παρέμβουμε. Ε, ανέκυψαν δυσκολίες και μπορώ να τις καταλάβω, αλλά δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όταν υπάρχουν τέτοιες αμφισημίες ή προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο ε, επιλογής των προγραμμάτων, ε, παρά την αυτονομία, την ανεξαρτησία της κριτικής επιτροπής, δεν πρέπει να απαντούμε πούμε, ε, ε, απεκδίοντας κάθε ευθύνη. Θα, δεν θα ήθελα αυτό να αποτελέσει πρόβλημα για μια μελλοντική επιλογή διότι προφανέστατα όλοι οι εταίροι μας θα παρακολουθούν ε, από κοντά τις εξελίξεις παρά είναι ξαναλέω νεόκοπος ο οργανισμός για να λειτουργεί έτσι και δεν πρέπει να επιτρέπεται να δημιουργούνται τέτοιου είδους αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή των προγραμμάτων και όχι αμφιβολία, είναι... Ε, ε, ε, δεν πρέπει να δημιουργείται πρόβλημα με την και αμφισβήτηση της επιλογής. Ενημέρωσα τον πρόεδρο και στην απάντηση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου έλεγε ότι είναι ανεξάρτητο το κέντρο και ότι δεν εμπλέκεται στις αποφάσεις της Κρητικής Επιτροπής. Αυτά για το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Ναι, μεν είναι ανεξάρτητο, αλλά πιστεύω ότι σε όλη αυτή την περιπέτεια ε, υπάρχουν πολλά μελανά σημεία και θα ήθελα να με καθησυχάσετε για το μέλλον ουσιαστικά. Paul Rübig, letzte Wortmeldung und dann müssen wir schauen, wie wir die Antworten hinkriegen. Ε, Επόμενος, και μετά θα πρέπει να κάνουμε και καμία απάντηση γιατί και μισή συνεχίζουμε με άλλο θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ για την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Ινστιτούτου γιατί αναφέρθηκαν και πολλές ε, δημιουργικές ιδέες. Το ερώτημά μου πηγαίνει προς την ε, κατεύθυνση της ε, περαιτέρω εκπαίδευσης τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και μπρο, καθώς ε, στην ίδρυση του Ιδρύματος στόχος μας ήταν, ε, ξέραμε ότι θα εργαστούμε με το 7ο πρόγραμμα, με όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτή η γνώση πώς θα μπορέσει να περάσει στο σύστημα εκπαίδευσης, στα πανεπιστήμια, στους καθηγητές, στους καθηγητές στη μέση εκπαίδευση μέχρι τα νηπιαγωγεία πώς θα πάει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα μεταφερθεί στα κλάστερ. Πρέπει να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί όλη αυτή η γνώση. Και βεβαίως μου άρεσε ε, αυτό το οποίο είπατε στην παρουσίαση, να έχουμε και τέλος αποτελέσματα για τους πολίτες, ε, τους πολίτες. Αυτό πάντα ονειρεύονταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι ο πιο ανταγωνιστικός χώρος του πλανήτη. Αυτή είναι η αποστολή δική σας, δηλαδή αυτό το οποίο ξέρουμε που βρίσκεται στα αρχεία και μαζεύει σκόνη και μίκητες Πώς θα απελευθερωθεί αυτό το δυναμικό. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να βρεθεί σωστές μηχανές αναζήτησης στους ενδιαφερόμενους πολίτες για να είναι με την τελευταία λέξη της, ε, της γνώσης. Δεν ανάγκη να μένουν αυτά τα πράγματα στο... στο πανεπιστήμιο, ούτε καν και μέσα στο πανεπιστήμιο. Βλέπουμε πως καθηγητής ε, συχνά διδάσκει αυτά τα οποία είχε διδαχθεί ο ίδιος τότε στο πανεπιστήμιο 30 χρόνια πριν. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα άτομα τα οποία διδάσκουν. Πώς θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο, να μεταφέρουμε τη γνώση που είναι διαθέσιμη σε πάρα πολύ λίγους να την κάνουμε χρήσιμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας προσπαθήσουμε τώρα να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Ο κύριος Ντεμπρούν θα δώσει πρώτα κάποιες απαντήσεις για τα γενικές ερωτήσεις και μετά αναλόγως με το ποιος θεωρεί ότι τον αφορά η ερώτηση ε, θα μου κάνει νόημα για να απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει και μισή σταματάμε για να περάσουμε και στα επόμενα σημεία. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ομαδοποιήσω ορισμένες ερωτήσεις που μας απευθύνατε ε, ως προς τα ερωτήματα της κυρίας Καρβάλιο για την ανεξαρτησία του Ινστιτούτου και την ε, πείρα μας σε αυτό το τομέα με βάση τα δεδομένα και της Κομισιόν θα ήθελα να σας πω ότι το Ινστιτούτο θα γίνει αυτόνομο. Προβλέπεται και η χρηματοδοτική του, χρηματοοικονομική του αυτονομία, η οποία θα αρχίζει στις 21 Ιουνίου. Όμως δεν θα είναι ανεξάρτητος οργανισμός, δηλαδή θα δρά από κοινού άλλους φορείς. Δηλαδή θα υπάρχει αλληλεξάρτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δείτε τον τομέα της εκπαίδευσης, αυτό είναι κάτι το οποίο απασχόλησε την Επιτροπή ως προς τη γνώση και την εμπειρία και το EIT ε, δεν θα ήταν αποδοτικό εάν υπάρχει επικάλυψη ικανοτήτων. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη δηλαδή ε, διαμόρφωση στοιχείων έτσι ώστε να έχουμε κοινή πλεύση. Ως προς τις συμβάσεις, την υπογραφή συμβάσεων, έχει μεγάλη σημασία να συνδέσουμε αυτό το ζήτημα με αυτό που είπε και η κυρία Ριέιρα σε σχέση με την έδρα των ΚΙΚΣ, τι λειτουργήσε και τι όχι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Ε, κάτι καταφέραμε, καταφέραμε κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν, διότι κάναμε αλλεπάλληλες δοκιμές. Οι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας επεξήγησαν για το πώς ε, λειτουργούν και έχετε αυτά αποτελέσματα όμως και το Ινστιτούτο δεν έχει επανδρωθεί πλήρως. Άρα μαζί με τα ΚΙΚΣ προσπαθούμε να προτρέξουμε κάπως έτσι ώστε να βρίσκονται επιτάπητος και όπως ξέρουν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι εκτελεστικοί διευθυντές, αυτό δεν είναι μία απλή διεργασία. Στη συνέχεια υπήρχε το θέμα της διάσκεψης των εμπλεκομένων φορέων ε, κατά πόσο επήλθε συμφωνία. Όπως σας είπα, το Ινστιτούτο άρχισε τη συζήτηση με τις θεματικές ενότητες για τα ΚΙΚΣ. Τα ε, παραδείγματα ε, αφορούν τον τομέα της υγείας, την γύρανση του πληθυσμού και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα που θα προσδιορίσουν τις δραστηριότητές μας. Υπάρχει μία ανοιχτή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ερχόμαστε σε διαβούλευση και με το κοινό και στο τέλος πιστεύουμε ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφανθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρούμε θεματικές ενότητες που θα απασχολήσουν τις ε, κοινότητες γνώσης. Δηλαδή θα συνδυάσουμε την έρευνα, την επιχείρηση και την εκπαίδευση για να ε, δώσουμε μια προστιθέμενη αξία. Ως προς τη συμμετοχή της βιομηχανίας στα ΚΙΚΣ θα ήθελα να πω ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε τα στοιχεία του 2010 ως προς την ανταγωνιστικότητα. Έχει αυξηθεί η συμμετοχή των βιομηχανιών. Είδατε και τον κατάλογο των εταίρων σε μια διαφάνεια. Ε, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής έτσι ώστε να υπογραφούν οι συμβάσεις και έκτοτε γνωρίζουμε ότι αυξήθηκε η συμμετοχή της βιομηχανίας το θέμα των ρίξ θα το αφήσω σε σένα, Μέρη. Η κυρία Μακής ρώτησε πώς ε, το θέμα των ε, εταιρικών σχέσεων και των καινοτομιών διασυνδέεται. Διότι ε, προσπαθούμε να βρούμε το δρόμο μας κι εμείς και να ορίσουμε το ρόλο μας για το μέλλον. Όμως το Ινστιτούτο ε, δεν μπορεί να βρίσκεται μόνο του στην έρημα εκτός όλων των άλλων μέσων, διότι έτσι θα πάψει να λειτουργεί. Θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη εικόνα έτσι ώστε να δώσει προστιθέμενη αξία και σε άλλα προγράμματα. Εδώ αναφέρομαι στα διαρθρωτικά ταμεία και γνωρίζω ότι και τα άλλα δύο κύκς, οι άλλες δύο κοινότητες γνώσης και καινοτομίας θα πρέπει να εξασφαλίσουν το πρόγραμμα που εντάσσουν στα προγράμματα εργασίας που αποτελεί το 75% του προϋπολογισμού έτσι ώστε να υπάρχουν ε, συνέπειες που να δράσουν ως καταλήξεις με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου. Στη συνέχεια το ερώτημα της κυρίας Έιλερ σε σχέση με την αποτίμηση των διαρθρώσεων. Είχαμε μία επταετή εταιρική συμφωνία και αυτό το θέμα μας απασχόλησε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Και φτάσαμε σε αυτά συμπεράσματα. Το Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο δεν θα ήθελε απλώς να δει ποιες προσπάθειες καταβάλλονται να ελέγχει τα έξοδα και μετά να καταβάλει τις πληρωμές. Θέλουμε αποτελέσματα και με βάση τα αποτελέσματα θα αποφασίσουμε για το νέο πολιετές πλαίσιο επενδύσεων. Τα αποτελέσματα αυτά θα θέλαμε να τα δούμε μέσα στα πλαίσια των KPI που χρησιμοποιούν τα KICS για να δούμε ποιες θέσεις εργασίας, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούνται, να δούμε αυτά τα βαθμολόγια και να δούμε τι ακριβώς μπορεί να γίνει έτσι ώστε να αποδώσουν οι επενδύσεις και τα χρήματα των φορολογμένων. Και αυτό που έχει σημασία είναι να γίνει μια συνολική αξιολόγηση. Βεβαίως ε, σημασία έχει και η εργασία του ίδιου του Ινστιτούτου που θα ενταχθεί σε αυτή την ε, αξιολόγηση. Τέλος, η κυρία Φαμπρέμπτ έθιξε ένα... Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε ο κύριος. Η κυρία Τράουτμαν κυρία Τράουτμαν. Πράγματι, θίγησαν ε, ερωτηματικά, υπήρξαν ερωτηματικά ως προς την επιλογή των ΚΙΚΣ και ο διαμεσολαβητής ζήτησε ορισμένες επεξηγήσεις. Τώρα εξαρτάται από τον διαμεσολαβητή να κάνει μία περαιτέρω αποτίμηση και να επανέλθει σε εμά αν χρειαστεί να επιληθεί το ολοζήτημα. Αυτά μπορώ να σας ε, πω, Πρόεδρε, επί του παρόντος. Ναι, έχετε το λόγο και εσείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στο ερώτημα για το ΡΙΚ και τα κέντρα συστέγασης. Τα κέντρα εκεί συστέγασης ε, είναι στη βορειοδυτική Ευρώπη. Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία και Γερμανία. Τα επιλέξαμε εκεί γιατί αυτά ήταν τα κέντρα που είχαν την υποδομή για συστέγαση που μπορούσαν να έχουν αυτό το οικοσύστημα εάν θέλετε για να υπάρχει στήριξη επιχειρηματική των ανθρώπων είχαν υποστηρικτικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, αλλά επιλέξαμε μετά εσκεμένα διαφορετική δομή για περιφερειακά κέντρα καινοτομίας, ε, τέσσερα από τα οποία δεν είναι στη Δυτική Ευρώπη, αυτά είναι στην Πολωνία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία και υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο και διαφορετικό εκεί που είναι η πρόσβαση στην τοπική κοινωνία και πληροφορίες για το τι χρειάζεται τοπικά στην Ευρώπη και βεβαίως και τη δυνατότητα να ε, το δώσουμε και εμείς αυτό. Και βεβαίως δεν θέλουμε κι εμείς να επεκταθούμε πάρα πολύ γρήγορα, θέλουμε να έχουμε συνεργασίες, αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε να σταθεροποιηθούμε ως νέα δομή, αλλά βλέπω πως θα εξελιχθούν τα πράγματα και θέλουμε να εμπλακούν και άλλες περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε υπήρχε ένα πολύ ε, ισχυρό σκεπτικό γι' αυτό. Αλλά αναφερθώ για το πρόγραμμα πλαίσιο 7 Κοιτάξτε, στο δικό μας ε, το πρόγραμμα περί κλίματος υπάρχει ήδη αρκετή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα πλαίσιο 7, οπότε ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Επίσης, στη... στις 17 Μαρτίου, όταν ήρθαν τα τρία κίκ στις Βρυξέλλες και συναντηθήκαμε με διαφορετικούς γενικούς διευθυντές, εμείς περάσαμε ένα ωραιότατο απόγευμα με πολλούς διευθυντές και το συμπέρασμα ήταν πώς θα είχαμε ξεχωριστά εργαστήρια και με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας για να δούμε τα κενά ε, μεταξύ του τι έκαναν ε, στο πρόγραμμα ε, πλαίσιο 7 και πού μπορούσαμε να συμπληρώσουμε και εμείς την προστιθέμενή μας αξία. Και τέλος βεβαίως στην ε, πράξη το μήνυμα μεταφέρεται και οι φοιτητέ μας το μεταφέρουν και όλα τα ιδρύματά μας έχουν πάρα πολύ εκτεταμένα προγράμματα επαφής, μένα πάνε σε τοπικά σχολεία και θα τον ενσωματώσουμε αυτό και αυτό στο ΚΙΚ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ένα μόνο μήνυμα σε σχέση με το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο σε σχέση με το μέλλον. Ε, ήδη έχουμε δώσει, έχουμε δώσει στοιχεία για την πράσινη ε, βίβλο ως προς τις κοινότητες σε σχέση με την ε, ε, πράσινη ενέργεια να βασιστούμε στα αποτελέσματα και όχι στις προσπάθειες που καταβάλλονται. Το δεύτερο είναι να μην συγχαίουμε την απλούστευση με την ομοιογένεια. Υπάρχει ένας διαφορετικός ε, κύκλος ε, δράσης. Μιλάμε για απλούστευση και όχι για ομοιογένεια. Επίσης, ας κρίνουμε με βάση την αποδοτικότητα και ας κρατήσουμε μόνο τα σχέδια που είναι αποδοτικά και ας δούμε τι θα κάνουμε ως προς αυτά που δεν αποδίδουν. Πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε ξεχωριστά. Ορισμένα θέματα αφορούν την συμμετοχή της βιομηχανίας ε, και αυτό αφορά και τα ερωτήματά σας στο, ΤΕΧΝΟ στο Ινστιτούτο, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας είδαμε τι προσέγγιση μπορούμε να ακολουθήσουμε. Νομίζω όμως ότι στον τομέα της αυτονομίας και της απλούστευσης ορισμένα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Διαφορετικά δεν θα κινηθούμε τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε και έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει απλούστευση προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Σε σχέση με την εκπαίδευση, θα ήθελα να μιλήσω για τη σημασία της εκπαίδευσης. Ένα από τα ζητήματα που δεν επιτρέπουν στην τεχνολογία να μπει στην αγορά ε, ε, έγκυται στο γεγονός ότι δεν συμβαδίζει η εκπαίδευση Εάν όλα αποτύχουν, πολλές φορές λέμε στους ενδιαφερόμενους διαβάστε τις, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Θα πρέπει όμως ε, αυτή η ανάγνωση να γίνει από τα πριν. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η εκπαίδευση να εμπλακεί με την αγορά εργασίας και να μην παραμείνει στα πανεπιστήμια. βεβαίως βασιζόμαστε στις αλλεπάλληλες δοκιμές, στην προσέγγιση δοκιμής και σφάλματος. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τη φάση της οικοδόμησης. Και όταν γίνεται στη φάση της οικοδόμησης, τα πράγματα δεν είναι τέλεια αλλά πουθενά δεν είναι τέλεια τα πράγματα εκτός από τον παράδεισο. Και θα ήθελα να μην ε, πάω αμέσως εκεί. Θα ήθελα να μου μείνει λίγος χρόνος πριν από αυτό. Όταν ε, ήμουνα διευθύνων σύμβουλος της Φίλιπς ε, έλεγα ότι αν όλα τα προσκόμματα πρέπει να τα υπερβούμε τότε αμέσως τότε δεν θα φτάσουμε πουθενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου και κύριοι. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί αυτά τα οποία είπατε μίλησαν από μόνα τους και θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ πέρα και μας αφιερώσετε χρόνο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Κυρίε και κύριοι, περνάμε σημείο 10. Εκτελεστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και καλωσορίζουμε ε, κάποιες κυρίες και κυρίους και το Συμβούλιο Έρευνας βεβαίω έχει εξελιχθεί και συμβάλλει στην πολιτική. Έχουμε λοιπόν κάποιους καλεσμένους οποίους χαιρετίζω και έχουν διαφορετικές αποστολές και η καθηγήτρια η κυρία Νοβότνη ζήτησε να τονίσουμε τις διάφορες πτυχές, γι' αυτό μοιράσαμε το χρόνο ομιλίας και λογικά θα ξεκινήσει η κυρία Νοβότνη. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι τιμή μου που ξαναέρχομαι στην Επιτροπή σας. Η Επιτροπή σας ε, Ε, ενδιαφέρονταν για μας πριν ξεκινήσουμε καν, οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι εξετάζεται σήμερα το που βρισκόμαστε. Να σας υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Μιλάμε για μια φοβερή ε, αλλαγή πολιτικής. Για πρώτη φορά θα χρηματοδοτούσε ε, την πολιτική εχμής η Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσης, εμείς ε, χρηματοδοτούμε συγκεκριμένους μεμονωμένους ερευνητές που πιστεύουμε πως ξέρουν που είναι τα όρια της επιστήμης και η μόνη, μία και μόνη αρχή μας είναι η αριστεία. Η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ένα νομικό μέσον, διότι ο ανταγωνισμός ε, ενέκυψε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το πλαίσιο ανταγωνιστικής δράσης. Αρχίσαμε να λειτουργούμε από το 2007. Έκτοτε είχαμε οκτώ ε, ε, εκκλήσεις για εκδήλωση, προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι έξι ε, έχουν συμπληρωθεί. Είχαμε 20.000 προτάσεις και είχαμε και πολλούς υπότροφους. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ μαζί μας. Πρόκειται για νέους ερευνητές και αυτό θα ήθελα να το τονίσω, διότι μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε τους νέους ερευνητές, τους αριστούχους ερευνητές μας. Επίσης, ε, πέρσι όταν ανακοινώθηκαν τα βραβεία Νόμπελ, είδαμε ότι στη φυσική είχαμε ε, να κάνουμε με ένα νέο ο οποίος ε, είχε εργαστεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και εμείς τον είχαμε ε, το προσλάβει για να προωθήσει τη δραστηριότητά του. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να φτάσουμε σε ε, ε, ρηξικέλευθες ανακαλύψεις που αποτελούν απαράβατο όρο της καινοτομίας. Εάν μιλάμε λοιπόν για έρευνα και τεχνολογία, αν μιλάμε για καινοτομίες, θα πρέπει να εξεύρουμε τη σωστή βάση έτσι ώστε να έχουμε μία εμπροστοφυλακή, η οποία άρχισε την εργασία της δύο δεκαετίες πριν. Τώρα, τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας ε, δεν μας ε, ικανοποιούν. Δεν έχουμε αρκετές γυναίκες υποτρόφους. Έχουμε στοιχεία επιτυχίας με βάση ένα 26% αλλά στο υψηλότερο επίπεδο υποτρόφων έχουμε ένα 12% μόνο γυναικών. Και αυτή είναι η ποσοστιαία αναλογία ε, γυναικών καθηγητών σε επίπεδο Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να τα καταφέρουμε καλύτερα και γι' αυτό υπάρχει και ένα σχέδιο ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών. Επίσης ε, δεν προσελκύσαμε πολλούς υποτρόφους εκτός Ευρώπης. Θα θέλαμε η Ευρώπη να ε, είναι αρκετά δελεαστική για έρευνα πώς ισχύει για τις, Ήπρα μέχρι, για τις μέχρι τώρα και την Νοτιοανατολική Ασία. Θα θέλαμε και η Ευρώπη να βρει τη σωστή της θέση και τώρα προωθούμε μια στρατηγική διεθνοποίησης έτσι ώστε και εμείς να κατέχουμε τη σωστή θέση στην παγκόσμια σκακέρα. Χαιρόμαστε διότι οι υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχουν μία κατανομή ανά την Ευρώπη, αλλά δεν είναι ίση κατανομή. Υπάρχει ένα σχέδιο αριστείας. Η αριστεία προσελκύει την αριστεία. Έχουμε ένα 50% που αφορά συγκεκριμένα Ινστιτούτα, το άλλο 50% αφορά συγκεκριμένους φορείς και Ινστιτούτα και Ιδρύματα, τα οποία έχουν ανταγωνιστική σχέση μεταξύ τους. Αυτό είναι το διαρθρωτικό πλαίσιο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δράση της νέας γενιάς έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία που να είναι συναρπαστική στο πενταετές αυτό πλαίσιο για να αναπτύξουν τις ιδέες τους και επίσης θα ήθελα να πω ότι για αυτή τη γενιά θα πρέπει να υπάρχει επιστημονική ανεξαρτησία πολύ νωρίτερα από ό,τι ίσχυε μέχρι τούδε στην Ευρώπη. Θα πρέπει οι νέοι να μπορούν να προωθούν όχι αυτό που επιθυμεί ο καθηγητής τους, αλλά αυτό που επιθυμούν οι, ίδιοι. Σε σχέση με τη, του, τα, τα Ιδρύματα Φιλοξενίας, Υπάρχουν θετικές επιπτώσεις που βλέπουμε στα πλαίσια αυτών των Ινστιτούτων. Επίσης, η ε, βιομηχανία κατανοεί πολύ καλά την αξία της έρευνας εμπροστοφυλακής. Γιατί διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει αριστεία, δεν θα υπάρχουν και νέα προγράμματα. Και ο βασικός μας στόχος είναι και η βιομηχανία να επιλέξει τις καλύτερες ιδέες και να τις αναπτύξει περαιτέρω μέσα στα πλαίσια του δρόμου προς την ε, καινοτομία. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας δεν έχει πρότυπα αξιολόγησης. Ορισμένα κράτη έχουν ε, αλλάξει τα συστήματα αποτίμησης και αξιολόγησης έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι πιο ανταγωνιστική. Επίσης, πρόσφατα προσθέσαμε δύο άλλα προγράμματα μικρότερης εμβέλειας. Βρισκόμαστε σε φάση δοκιμής, δοκιμών. Πρόκειται για, μια, για ένα πολύ μικρό μερίδιο του προϋπολογισμού και βεβαίως ελέγχουμε ε, εκ του σύνεγγι αποτελέσματα. Προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε εκείνους που εργάζονται ε, με βάση νέες ιδέες έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο υπάρχει μια νέα συλλογιστική ή ενηλογική βάση για τη σύσταση επιχειρήσεων έτσι ώστε να υπάρχει ε, παροχή κεφαλαίων για να δούμε κατά πόσο, πώς μάλλον έχει η έκβαση αυτών των νέων έννοιων. Επίσης, ε, το σχέδιο υποτροφιών συνεργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτές τις υποτροφίες σε ε, δύο με τέσσερις βασικούς ερευνητές με βάση την ε, ανάντη προσέγγιση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι συνδέοντας αυτή την ε, ε, αυτή τη διαδικασία συνέργειας με δύο τέσσερις βασικούς ερευνητές θα μπορέσουμε να διανοίξουμε νέες οδούς συνεργειών ή ε, σύγκληση όπως την κατονομάζουν οι Αμερικανοί. Προς το τέλος θα ήθελα να αποστείλω ένα βασικό μήνυμα και θα ήθελα να πω ότι πάντα υπάρχει ε, χώρος στην κορυφή. Εάν δηλαδή Ε, υπάρχει ο ίδιος ε, ενθουσιασμός από τους υποτρόφους όταν δούμε πώς αλλάζει αυτό το πλαίσιο και η εικόνα βλέπουμε ότι υπάρχει σωστή άμυλα μεταξύ τους σε αυτό το επιστημονικό περιβάλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ζήτηση στη νέα γενιά έχουμε ένα 42% αύξηση στις αιτήσει, ιδιαίτερα στην φυσική, ε, την μηχανική, χημεία, αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην κοινωνιολογία. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση λοιπόν στις αιτήσει για υποτροφία και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι υπάρχει πολύ υψηλή ποιότητα, η οποία παραμένει πολύ υψηλή. Γι' αυτό θεωρούμε ότι υπάρχει χώρος στο υψηλότερο σημείο, στο επίπεδο των αριστούχων. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μία, ένα ποσοστό χαμηλής επιτυχίας, ένα δείκτη 13,8% σε σχέση με τους ε, τελευταίους πέντε διαγωνισμούς και θα θέλαμε να προσελκύσουμε και νέους ερευνητές υψηλών προδιαγραφών εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρώπης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μέσω πρόθεσμα οι χώρες που δεν τα κατάφερναν πολύ καλά τον, ε, το τελευταίο διάστημα θα έχουν υψηλότερη ε, αναλογία, έναν υψηλότερο δείκτη. Ο Πάμπλο θα σας ε, μιλήσει και για τον φορέα ο οποίος ασχολήθηκε με αυτή την ροή εργασίας που, η οποία ανέρχεται στο 3,5% όπως βλέπουμε από τα διοικητικά έξοδα. Ως προς αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο μπορώ να σας ε, μιλήσω ε, για τις πέντε συστάσεις του εγγράφου προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να παραμείνουμε στο επίπεδο της αριστείας. αυτό είναι το κλειδί επιτυχίας για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και για την εμπροστοφυλακή μας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μία αναθεώρηση, ένα σύστημα αναθεώρησης μεταξύ ομοτήμων και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι επιλέγουμε το πάνελ ανάμεσα στα καλύτερα στοιχεία. Μιλάμε για πλούστευση διεργασιών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ενιαίες προδιαγραφές και όταν υπάρχουν κράτη ή περιφέρειες που υπολειτουργούν ή που αποδίδουν, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε με ένα δημιουργικό περιβάλλον για την έρευνα και την ανάπτυξη. Ναι, κοιτάξτε τώρα βλέπουμε πως ο χρόνος πιάζει, πιέζει και θα πρέπει να βιαστούμε λίγο όλοι, αλλιώς θα μπορέσουν να ρωτήσουν και όλες οι συνάδελφοι κύριος Αμόρ θα μας πει λίγα ακόμα πράγματα για την εκτελεστική υπηρεσία. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βασικό μου μήνυμα σήμερα είναι ότι η καθηγήτρια Χαλκιανόρτη μα μας ε, περιέγραψε τι προσπάθειες που έχουν γίνει, δηλαδή επιλογή των βελτίστων ιδεών, προώθησή τους, δημιουργία ευνοϊκού κλίματος ε, για έρευνα, αλλά χρειάζεται και επιμελητία, ε, γραμματιακή, πέρα από την έρευνα. Έχουμε τους στόχους της αριστείας και θα ήθελα να προσπαθήσω με την παρουσίασή μου να σας πείσω ε, για το ότι ασχολούμαστε και με την αριστεία και με τη διοίκηση και με την ποταπή γραφειοκρατία. Ναι, ναι, μου το είπατε και θα το σεβαστώ. Πρέπει να είμαι σύντομο, θα μιλήσω πιο γρήγορα. Ε, για να σας δώσω λίγο το ιστορικό υπόβαθρο, να σας πω ποιο είναι το μέγεθος του Συμβουλίου στα πλαίσια του ε, ευρύτερου προγράμματος. 15% ε, του προϋπολογισμού, αυτό είναι το δικό μας τμήμα περίπου. Αρχίσαμε με μόνο 300 εκατομμύρια και γρήγορα αυξήθηκαν τα ποσά και στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο θα έχουμε το μεγαλύτερο τμήμα των κονδυλίων 1,8 δί το χρόνο. αυτό θα είναι ο προπολογισμό μας και θα αναλάβουμε τις μεγαλύτερες προσκλήσει για υποβολή προσφορών του προγράμματος ε, πλαίσιο. Θα ήθελα να εξηγήσω λίγο ποιο είναι το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για όσου δεν το γνωρίζουν. Έχουμε δύο είδη υποτροφίων. Ε, το, η μία κατηγορία δίνεται στην αρχή αρχικές επιδοτήσεις, αρχικές υποτροφίες και οι προχωρημένες. Αυτό το μοντέλο το χρησιμοποιούσαμε εξ αρχής και βλέπετε ότι για την πρώτη κατηγορία το προπολογισμό είναι περίπου 2 εκατομμύρια για πενταετή περίοδο και ε, κατά τι αυξημένο το ποσό 3,5 εκατομμύρια για 5 χρόνια για τις ε, προχωρημένε προχωρημένες ε, επιδοτήσεις, υποτροφίες. Ούτως ή άλλως όταν μιλάμε για ανθρώπους που κάνουν διδακτορικό πρέπει να φτάσουν στα 27, 28. For, for grants, which also Τώρα, ε, σας μίλησα για τη διοίκηση και την αποτίμηση. Νομίζω ότι έχουμε καλές επιδόσεις. Έχουμε την, τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της ζήτησης που προβλέπουμε για τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για τη διοικητική διάσταση των πραγμάτων και ξέρω ότι σε τέτοιους χώρους ε, είναι πολύ συζητημένα τα θέματα της απλούστευσης, ε, της επίσπευσης της χορήγησης των ε, υποτροφιών κτλ. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι βεβαίως της πρόσκλησης υποβολής προσφορών παρότι έχουμε μεγάλο κομμάτι του προγράμματος πλαισίου και ε, η συνήθις ε, περίοδος ε, για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι 14 έως 20 μέρες. Είναι κάτι το απίστευτο. Οι τράπεζες χρειάζονται μόνο 2-3 μέρες. Η υπότροφη είναι πολύ δημιουργική και μέσα σε διάστημα 10 ημερών πρέπει να, να προσδιορίσουμε τους κανόνες, να κανονίσουμε τις σχέσεις με την τράπεζα Uh, είναι ελαφρύ το διοικητικό μας άκθος και έτσι θέλουμε να παραμείνει. Είναι απλό το μοντέλο λειτουργίας μας ε, και η δομή μας δεν είναι τόσο παλιά. Καταλαβαίνετε ότι η επιστημ... το Επιστημονικό Συμβούλιο κάνει την επιλογή, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί για αυτή την πενταετία κάθε πρόγραμμα και μεριμνάστε διοικητικός πώς να τηρούνται οι κανόνες, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υποστηρίζει το τμήμα που ασχολείται με τα διοικητικά ζητήματα. Το προσωπικό μας, ε, ε, περίπου 330 άτομα έχουμε και δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε τους 389 μέχρι το πέρας του προγράμματος πλαίσιο και βλέπετε κυρίως έχουμε συμβασιούχους, έχουμε βέβαια και κάποιες προσωρινές ε, συμβάσεις κυρίως για τους επιστημονικούς αξιωματούχους, άνθρωποι κυρίως με τις απαιτούμενες γνώσεις και τα διδακτορικά για να είναι στη θέση να παρακολουθούν τις εξαιρετικές προτάσεις για τις οποίες χορηγούμε τις υποτροφίες. Ε, θα ήθελα τώρα να σας δείξω ε, ένα βασικό ε, αριθμητικό στοιχείο, δηλαδή ο λειτουργικός προϋπολογισμός του οργανισμού 2,5% είναι το διοικητικό κομμάτι στον λειτουργικό μας προϋπολογισμό, 2,58% πιο συγκεκριμένα. Ε, μπορείτε να κάνετε ένα παραλληλισμό με άλλα αντίστοιχα κέντρα, δηλαδή ποιο κομμάτι του προϋπολογισμού τους αφιερώνουν στα διοικητικά. Ε, δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα παρόλα αυτά να αναφερθώ σε τρεις βασικές ε, ιδέες. Προσπαθ... Επιδιώκουμε την απλούστευση και κάνουμε πειράματα με αυτά τα προγράμματα και νομίζουμε ότι μπορούμε να απλοποιήσουμε περαιτέρω το ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Επίσης, ε, ε, για τη διοίκησή μας αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αντιμετώπιση των εταίρων μας. Εάν υπάρχουν κάποιες ανησυχίες προσπαθούμε να μάθουμε από τα λάθη μας, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την, ε, τις σχέσεις που έχουμε με τους εταίρους μας. Είναι μια διαρκή προσπάθεια. Τελευταία ιδέα, ο Παφ Ντάντι που είναι ένας ράπερ, ε, αναφέρθηκε στο Notorious Big ε, ε, και του είπε μην αλλάξεις ε, το έγγραφο, άλλαξε το όνειρο και εμείς αυτό κάνουμε. Δεν θέλουμε να τροποποιούμε τη διαδικασία, θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα νέο όνειρο. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την κυρία Μονιέ. Ελπίζω να προέφερα στο δαρμά σας. Όχι. Να το πρώτο λάθος ήδη. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θα μας πείτε γιατί είναι χρήστης του προγράμματος και μπορεί να μας διηγηθεί ποια αποτελέσματα υπάρχουν στον τομέα της. Οπότε έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να σας πω πως χρησιμοποιήσαμε αυτά τα υπέροχα λεφτά, τα πολλά λεφτά που μας έδωσαν. Το εργαστήριό μου ε, εργάζεται πάνω στη μνήμη και ήδη από την αρχαιότητα, από το Μεσαίωνα βλέπουμε πως υπήρχαν διάφορα μνημονικά κόλπα για να, μαθαίνει ο κόσμος κάποια πράγματα. Βλέπετε εδώ πέρα με το να βάζει κάτι σε συγκεκριμένο σημείο ε, όπως ε, το χέρι του Γκουίντο Νταρέτσο εδώ πέρα βλέπετε που αντιστοιχούσε κάποια πράγματα στα δάκτυλά του και βεβαίως αυτό φαίνεται και στο έργο του Μποτιτσέλη ο οποίος μας δείχνει τη θεία κομμωδία του Δάντη. Ο Δάντης κατεβαίνει στην ε, κόλαση και τους βλέ... βλέπει τον κόσμο σε διαφορετικά μέρη και άρα τους κατανέμει στους 7 κύκλους της κολάσεως για να θυμάται που είδε τον, κανένα, τον καθένα. Οπότε έτσι λειτουργεί λοιπόν η μνήμη. Οπότε εμείς εργαζόμαστε στην μνήμη σε σχέση με τον χώρο. Βλέπετε το σκίτσο αυτό εδώ πέρα, τον ε, υπόκαμπο εδώ πέρα με κίτρινο χρώμα. Αυτή είναι η δομή η οποία θα σας επιτρέψει ε, να θυμάστε τα πράγματα τα οποία σας είπα, εάν θυμάστε τίποτα, θα έχουν αποθηκευτεί σε κάποια κύτταρα του υποκάμπου και μετά μεταφέρονται αλλού στον εγκέφαλο. Αυτό ήταν γνωστό από τη δεκαετία του 1950 όταν ε, εγχειρίστηκε ο ασθενής HM γιατί υπέφερε από επιληψία. Όταν, όταν αφαιρέθηκαν οι υπόκαμποι, κάτι το οποίο γίνεται ακόμα και σήμερα, ο ασθενής αυτός δεν μπορούσε να έχει πλέον νέες αναμνήσεις. Όλες του οι παλαιές αναμνήσεις υπήρχαν, θυμόταν τα παιδικά του χρόνια, επεισόδια από τα, βρεφικά, από τα παιδικά του χρόνια, αλλά δεν μπορούσε να σχηματίσει νέες αναμνήσεις. Έτσι διαφοροποιούμε και σε μοντέλα με πειραματόζωα, με το να επηρεάζουμε τον υπόκαμπο, που επηρεάζουμε μόνο τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και αφήνοντας εκτός την μακροπρόθεσμη μνήμη. Από το 1950 λοιπόν γνωρίζουμε πως υπάρχουν διαφορετικά είδη μνήμη σε διαφορετικά σημεία του εγκεφάλου και το δικό μου το εργαστήριο ασχολείται με αυτή τη συγκεκριμένη δομή. Τώρα, η μνήμη ή χωρική, εάν θέλετε κανείς να, αν θέλετε να θυμάστε πως πάτε από εδώ στο τρένο, εάν βάλουμε ηλεκτρόδια στον ε, υπόκαμπο, είναι, είναι δύσκολο εδώ πέρα να χειριστώ το λέιζερ, είναι αυτό το μπανανοειδές σχήμα στον εγκέφαλο του ποντικού, όπως και στον ανθρώπου άλλωστε. Και εάν εργάζεται σε ένα κουτί, σε ένα λαβύρινθο ο ποντικός και γεμίσουμε την, ε, και κυρματογραφήσουμε την πορεία του, βλέπετε τη φοβερή ανακάλυψη του Τζον Οκίφ, η τροχιά δηλαδή που ακολουθεί το ποντίκι. Με μαύρο βλέπετε την τροχιά και με κόκκινο βλέπετε ένα συγκεκριμένο κύτταρο, ένα νευρώνα που κινητοποιείται κάθε φορά που βρίσκεται σε συγκεκριμένο μέρος το ποντίκι. Οπότε χαρτογραφούμε το περιβάλλον μας με αυτά τα τοπικά κύτταρα κάθε φορά που βρίσκεται κάποιος σε ένα σημείο και κάθε φορά που το ποντίκι βρίσκεται σε αυτό το κουτί θα χτυπήσει σε ένα μόνο σημείο αυτό το κύτταρο. Αυτά τα κύτταρα τα τοπικά λοιπόν χαρτογραφούν το χορτό εργαστήριό μου όμως ενδιαφέρεται όχι μόνο για αυτά τα τοπικά κύτταρα τα οποία τα βλέπετε δεξιά με κόκκινο αλλά και για τα μεμονωμένα γαλάζια κύτταρα είναι εκείνα τα α, κύτταρα γκάμπα τα λεγόμενα τα οποία μου έδωσε λεφτά μου έδωσαν λεφτά για να εργυνήσω, τα οποία είναι, αν θέλετε, οι διευθυντέ ορχήστρας Τα κόκκινα κύτταρα, τα τοπικά είναι αυτά τα οποία παίζουν τη μουσική, αλλά τα μπλε κύτταρα είναι αυτά τα οποία συγχρονίζουν τα μπλε κύτταρα για το πότε θα κινητοποιηθούν για να έχουμε μια αναπαράσταση του χώρου στο μυαλό μας. Θα περάσω αυτή τη διαφάνεια. Οπότε βλέπετε ε, προσπαθούμε να δούμε ποια μόρια κινητοποιούνται και δημιουργούμε κάποια μοντέλα και το βάζουμε σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια, αλλάζοντας κάποια μόρια για να μην μπορούν να δουλέψουν συγχρονισμένα οι διευθυντές αυτή η ορχήστρα στο είδος κυτάρων που σας είπα. Οπότε πάμε από το μόριο στο κύτταρο, στα δίκτυα, στο μοντέλο του δικτύου και αλλάζουμε μέσω γενετικών μοντέλων συγκεκριμένα από τα κύτταρα διευθυντών ορχήστρων, ορχήστρα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ακριβώς τα μπλε αυτά κύτταρα πως ε, αυτά τα διευθυντικά θα λέγαμε κύτταρα είναι μόνο ένα 10% των ευρικών σας κυτάρων και ε, έχουν εδώ πέρα μία συγκεκριμένη δίωδο της, ε, την οποία τους αφαιρούμε για να μην μπορούν να κινητοποιηθούν συγχρονισμένα και τότε δοκιμάζουμε στα ποντίκια μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη μνήμη. Πώς γίνεται αυτό με τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Τους βάζουμε σε ένα λαβύρινθο και στην άλλη άκρη έχει λίγο ζαχαρούχο γάλα. Και κάθε φορά που πρέπει να ξεκινήσει στο σημείο Α ή στο σημείο Β, κάθε λίγες μέρες, σε λίγες μέρες θα μάθει πώς βρίσκεται, βλέπετε εκεί, στο σημείο Γ το ζαχαρούχο γάλα. Θα το θυμάται αυτό για εβδομάδες και μήνες το ποντίκι. Γι' αυτό μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Βλέπετε πως το ποντίκι ε, κάνει αρκετά λάθη, ένα 50%. Αλλά όπως περνάει ο χρόνος, ε, είτε το, στο α είτε στο β το βάλουμε, θα πάει κατευθείαν στο ζαχαρούχο γάλα. Μετά, η βραχυπρόθεσμη μνήμη που είναι π.χ. Ε, να θυμόμαστε ένα αριθμό τηλεφώνου μέχρι να τον πληκτρολογήσουμε, αλλά όχι την επόμενη μέρα εάν δεν το επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, τη δοκιμάζουμε ως εξής, τα βλέπετε στα δεξιά. Μπαίνει σε έναν λαβύρινθο σχήματο ταφ, ποντίκι, δεξιά υπάρχει ζαχαρούχο γάλα, μετά το βάζουμε πίσω στην αρχή, ανοίγει αυτό το κομμάτι που ήταν κλειστό και τώρα υπάρχει μία νέα μορφή, οπότε λειτουργούν σαν τους ανθρώπους τα ποντίκια, τους αρέσει η καινοτομία. Εάν έχει πάει στο δεξί κομμάτι θα πάνε συνέχεια στο καινούργιο και για να θυμάται ότι έχει πάει στα δεξί κομμάτι πρέπει να έχουν κάποιο είδους βραχυπρόθεσμη μνήμη. Και πάλι αφαιρώντας αυτά τα μόρια που κάνουν τα κύτταρα αυτά να λειτουργούν συγχρονισμένα, δεν λειτουργούν ε, εξίσου καλά τα ποντίκια, όπως βλέπετε και στο διάγραμμα μιλάμε ε, ότι έχουν ένα 90 με 100% ακρίβεια, ενώ τα μεταλλαγμένα στα οποία δεν υπάρχει αυτό το μόριο έχουν πολύ χαμηλότερη απόδοση. Έχουμε λοιπόν τα τοπικά αυτά κύτταρα. Αυτά εδώ πέρα τα έχουμε κάνει όπως σας είπα με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και βλέπετε πως ε, κάνει βόλτα στο ποντίκι και βλέπετε πως ε, αυτό το κύτταρο θα κινητοποιηθεί όταν φτάσει εκεί και αυτό το κύτταρο όταν φτάσει αλλού και αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε μέρα συγκεκριμένο κύτταρο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση. Εάν πάρετε λοιπόν αυτά τα κύτταρα, τα, τους διευθυντές ορχήστας που λέγαμε, βλέπουμε πως ε, δεν είναι τόσο ακριβής ο προσανατολισμός. Οπότε δεν υπάρχει μία αναπαράσταση του χώρου όπως θα έπρεπε αυτή να είναι. Και Κάτι το οποίο επίσης αλλάζει όταν επανερχόμαστε την επόμενη μέρα. Κατά κανόνα αυτά τα τοπικά κύτταρα όπως βλέπετε στα αριστερά λίγες ώρες αργότερα σταθεροποιούνται ενώ στα μεταλλαγμένα ποντίκια είναι πιο μουτζουρωμένα όπως βλέπετε εκεί και εάν πάτε μία ώρα αργότερα δεν είναι σταθερά τα κύτταρα αυτά. Οπότε δεν υπάρχει η αναπαράσταση του χώρου και τα τοπικά αυτά κύτταρα δεν είναι σταθερά. Οπότε η ε, χωρική μνημή επηρεάζεται. Τέλος, να σας πω πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τα κύτταρα με ικές κατασκευές, να πάμε σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και να επηρεάσουμε μόνο τον υπόκαμπο, αφήνοντας όλο τον υπόλοιπο εγκέφαλο άθικτο και να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Αυτό ήταν επίτευγμα των τελευταίων ετών. Και τέλος, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, στην τελευταία διαφάνεια, αν έχουμε ένα ποντίκι εδώ πέρα ή αρουραίο, μπορούμε να βάλουμε οπτική ίνα στον εγκέφαλο και να ερεθίσουμε με μπλε φως και να ενεργοποιήσουμε μόνο τα κύτταρα αυτά και διευθυντές ε, ορχήστρας όπως τα είπα για να δούμε τι γίνεται ενώ κάνουμε αυτό το τεστ. Μπορούμε λοιπόν να χειριστούμε αυτά τα κύτταρα είτε γενετικά είτε να χειριστούμε τη δραστηριότητά τους ενεργοποιώντας μόνο τα κύτταρα αυτά διευθυντές με μπλε φως. Κατ' λοιπόν ε, η χρηματοδότηση που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα, εγώ και οι συναδελφοί μου, ήταν για να μελετήσουμε τη μνήμη τη μνήμη τη μελετάμε με το να αναμειχθούμε σε αυτά τα κύτταρα τα οποία χαρακτήρισα διευθυντέ ορχήστρες για να συγχρονίζουν μεγάλα σύνολα κυτάρων που έχουν μια αναπαράσταση του χώρου στον εγκέφαλο του ζώου και μπορούμε μετά να χειραγωγήσουμε τα ζώα και να δούμε πώς αλλάζει η απόδοσή τους. Έχω βάλει τα ονόματα τεσσάρων συναδέλφων, αλλά για να γίνουν αυτά τα πειράματα χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά. Έχω 25 άτομα στο εργαστήριό μου που εργάζονται πάνω σε αυτά τα θέματα. Επί 5 χρόνια μόνο για να φτιάξουμε το γενετικά τροποποιημένο ποντίκι χρειάζεται 1,5 έτος και οι μελίτες που έδειξα χρειάζονται 3 με 4 έτη. Οπότε χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, μεγάλες ομάδες, αφενός ηλεκτροφυσιολόγους και μοριακούς βιολόγους και επιστήμονες μελετούν τη συμπεριφορά. Οπότε πάμε από τα μόρια στην συμπεριφορά για να μελετήσουμε κάτι το οποίο δεν έχει σημασία προφανώς μόνο για τα ποντίκια. Οι ίδιες δομές, τα ίδια κύτταρα είναι και στον δικό μας εγκέφαλο και ε, ελπίζω να σας βοηθήσουν να θυμάστε αυτά τα οποία είπα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Äh, Ευχαριστούμε όχι μόνο για την ε, παρουσίαση αυτή, αλλά και για την ε, ένταση και για το ότι μας ε, παρουσιάσετε το τι, το τι γίνεται με τα χρήματα αυτά για να αποκτήσουμε μια αίσθηση. Δεν ξέρω μήπως με την αίθουσα αυτή μπορούμε να κάνουμε τους συναδέλφους να βρίσκουν τη σωστή αίθουσα όταν συνεδριάζουμε. Όχι, όχι, εντάξει. Αστειεύομαι. Λοιπόν, να δώσω τον λόγο στον Δόκτωρ Μίτια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντάχει, θα μιλήσω, θα δω τις διαφάνειες πολύ σύντομα και θα μιλήσω για το ρόλο της, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Νομίζω ότι υπήρχε μεγάλη πολιτική θέληση, δεν πρόκειτο για θαύμα. Το Επιστημονικό Συμβούλιο του ERC ε, εργάστηκε πολύ δραστήρια τη νομοθεσία του, προγράμμα, του 7ου προγράμματος πλαισίου θεωρήθηκε ότι με τη λήξη θα έχουμε ένα νέο μέσο και γι' αυτό υπάρχει ε, το Ανώτατο Συμβούλιο υπό την διοίκηση της κυρίας Φράιμπερκερ από τη Λετωνία και στη συνέχεια φτάσαμε σε ένα πρόγραμμα δράσης με στόχο αυτή η, διάρθρωση του ERC να είναι ιδιαίτερα εύρωστη και να μπορεί να συνεργαστεί με όλες τις ε, επιστημονικές κοινότητες του κόσμου. Με βάση αυτό το πρόγραμμα δράσης έχουμε μία μόνιμη επιτροπή που ασχολείται με την ανανέωση του Συμβουλίου Επίσης ε, βλέπουμε τις διοικητικές διαδικασίες, τις αναθεωρούμε, καθώς και τη διαδικασία αποτίμησης που έχει μεγάλη σημασία για να κρατήσουμε το επίπεδο αριστείας που επιθυμούμε. Λαμβάνουμε υπόψη και επεξεργαζόμαστε και τα νομοθετικά και νομικά κείμενα σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων. Άρα πρόκειται για ένα εργαστήρι, αν θέλετε, για νέες ιδέες, όπου εποάζουν οι νέες ιδέες. Υπήρξε και μία άλλη αναθεώρηση, το Συμβούλιο από Φανθήκε και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011 θα πρέπει να ελέγξει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και αυτό γίνεται την κατάλληλη χρονική στιγμή διότι προσπαθούμε να ε, συντάξουμε το νέο πρόγραμμα δράσης. Βλέπουμε ότι το ERC στέφθηκε από επιτυχία όλοι ομόφωνα θεώρησαν ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας είναι απότοκο μιας πολύ, καλή εφαρμογής, πολύ καλής εφαρμογής του 7ου προγράμματος ε, δράσης. Η κυρία Φράιμπεργκερ θα διασφαλίσει την συνέχεια αυτής της διαδικασίας εποπτείας. Και επίσης είδαμε ότι έχει επιτελεστεί ε, πραγματική πρόοδος και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και θέματα απλούστευσης μέσα στα πλαίσια του 7ου προγράμματος πλαισίου και στα πλαίσια της ε, διακυβέρνησης. Άρα ε, συστάθηκε η ομάδα εργασίας πέρσι. Θα δείτε και τον... Θα έρθετε σε επαφή και με τον πρόεδρο της Task Force και είχαμε και νομικές συμβουλές και πραγματογνωμοσύνη από την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Θα, έχουμε, θα φτάσουμε σε συμπεράσματα τον επόμενο μήνα για την πλήρη εφαρμογή του Εβδόμου πλαισίου. Βεβαίως, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει στεφθεί από επιτυχία διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αριστεία και αυτό θα πρέπει πάντα να μας απασχολεί. Αποτελεί απόλυτη ανάγκη. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα χωρίς αριστεία. Επίσης το ERC είναι ένας οργανισμός μάθησης και είδαμε ότι τα πρότυπά μας είναι ευανάγνωστα από όλους, εύκολα προσπελάσιμα και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα πρότυπο ε, διακυβέρνησης που εξασφαλίζει μεγάλη ε, αυτονομία. Πρέπει να βασιζόμαστε στην εμπιστοσύνη και το τέταρτο στοιχείο είναι μία ε, ανάντη προσέγγιση. Επίσης έχει σημασία οι επιπτώσεις, έχουν σημασία οι επιπτώσεις στα εθνικά συστήματα, έτσι ώστε να λειτουργεί το σύστημα σαν ε, μια ακτινογραφία για να δουν τα κράτη-μέλη τι πρέπει να επιτελέσουν, τι εργασία πρέπει να επιτελέσουν. Άρα όλα αυτά τα μαθήματα τα συνάγουμε και τα εντάσσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Πρόκειται για μια πραγματική επιτυχία και χαίρομαι διότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από την Κομισιόν θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συνεχίσουμε αυτή την επιτυχή μας πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν χρόνο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Κύριε Γιόρταν Σίσελη, Α, λίγο έτσι σύντομα τις ερωτήσεις, ε, για να τελειώσουμε και μισή, γιατί έχουμε και άλλα μετά. Ρωμάνα Γιόρνταν Σίσιλη. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα, για τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Νοβότνη. Ε, μας είπε ότι επιθυμεί να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που να συμμετέχουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός. Είδα τα έγγραφα τα οποία λάβαμε πριν από την παρουσίασή σας και βλέπω ότι υπάρχει υποεκπροσώπηση ορισμένων κρατών μελών και ορισμένα δεν εκπροσωπούνται καθόλου. Είπατε ότι ο λόγος είναι η αριστεία, η αναζήτηση της αριστείας. Θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε αξιολογήσει την κατάσταση, ποιοι είναι οι λόγοι και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα αποτελέσματα, πώς μπορούμε να αποτιμήσουμε τους ερευνητές από αυτές τις χώρες. Είπατε ότι υπάρχει χώρος. Δεν θα πρέπει να χάνουμε ορισμένα λαμπρά μυαλά από αυτές τις χώρες. Με εξέπληξε η παρουσίασή σας και τα, το τελικό σας συμπέρασμα. Είπατε δηλαδή ότι ό,τι ισχύει για τον εγκέφαλο των ποντικών ισχύει και για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να σας ευχαριστήσω για τις παρουσίες. Έλειπα στην αρχή βεβαίως γιατί ψηφίζαμε σε μια άλλη επιτροπή και πολλοί συνάδελφοι είχαν πρόβλημα και εγώ επίσης. Να ξεκινήσω με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Συγχαρητήρια σε όλους εξελίσσονται τα πράγματα. Εμένα θα με ενδιέφερε να μάθω το πώς βλέπετε τη μελλοντική εξέλιξη των ε, προγραμμάτων, την προώθηση της ε, έρευνας. Θα προωθήσετε με μονομένους ερευνητές ή συνεργασίες. Πρώτον δεύτερον, κυρία Νοβότνη, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε και η κυρία Σίσελη, η ανάλυση ε, έδειξε πως ε, κάποιες χώρες δεν συμμετέχουν καθόλου και αυτό ήταν συγκλονιστικό πραγματικά. Ποιες ήταν οι αιτίες ε, δεν ξέρω, ίσως να υπάρχουν εξαιρετικοί ερευνητές οι οποίοι όμως να πήγαν σε άλλες χώρες και εκεί να δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια και άρα να μην φαίνονται στα στατιστικά στοιχεία. Αλλά εάν μπορούσατε να να το δείξετε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, εσείς γιατί θεωρείτε, γιατί δεν υπάρχουν ε, συμμετοχές από κάποιες χώρες και ποιο, ε, ποια μέτρα θεωρείτε εσείς ότι μπορούν να ληφθούν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Τέλος, για το EIT, ε, δεν ξέρω αν ακούστηκε ήδη, αλλά είναι και το θέμα, όπως είπαμε, της μακροπρόθεσμας μνήμης. Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα μπορεί να επιδείξει ήδη το EIT υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και τι χρειάζεται βελτίωση στη δομή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Έρευνας. Ε, έχουν φύγει αυτοί. Έχουν φύγει από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας φύγαν ήδη. Ε, να θα το οργανώσουμε. Κρίστιαν Χέλλερ, πρώτα απ' όλα σας συγχαίρω Ξέρετε, μου δίνει μεγάλη χαρά το να έρχεστε από το συγκεκριμένο ίδρυμα με το οποίο και εγώ έχω μία σχέση. Εν πάση περιπτώσει, το... ο εγκέφαλος ε, του ποντικού που μας αναλύσατε μου θυμίζει βεβαίως τον πικρό αγώνα που δώσαμε για να υπενθυμίσουμε, για να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία του ERC και τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερο ερώτημα, τονίσατε πάρα πολλές φορές ε, το θέμα της αριστείας και αυτό ήταν κάτι το δύσκολο στο πρόγραμμα πλαίσιο 7. Τώρα έχουμε ε, κάτι το διαφορετικό. Κάνουμε μία διάκριση ε, από πλευράς σάρτιο, από πλευράς Κομισιόν ε, μεταξύ επιστημονικής καινοτομία, επιστημονικής αριστείας και αριστείας στην καινοτομία. Το, και βέβαια έχουμε ως κριτήριο επιλογή στην επιστημονική αριστεία και μετά έχουμε την διαφοροποίηση αυτή με την, με την αριστεία στην καινοτομία. Πόσο το βρίσκεται λογικό να γίνεται αυτή η διάκριση. Και βεβαίως το άλλο ερώτημα αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Έχουμε μια καμπύλη, βλέπετε στο πρόγραμμα πλαίσιο τα τελευταία δύο χρόνια εκταμιεύονται τα περισσότερα λεφτά σε ποιο βαθμό ξαναξεκινάει από το μηδέν αυτή η καμπύλη μετά το τέλος του προγράμματος, δηλαδή μηδενίζονται τα κονδύλια και ξαναρχίζουν και πώς θα μπορούσε να αυξηθεί, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Είναι σαφώς αυτός ο στόχος του Κοινοβουλίου, αλλά τεχνικά πόσο έχετε λάβει υπόψη αυτό το θέμα, ότι δηλαδή πάντα με τη λήξη του προγράμματος έχουμε τα δύο τελευταία χρόνια υψηλό επίπεδο και μετά τίποτα και χρειάζεται ξανά μια κινητοποίηση για να υπάρχει και μια συνέχεια, γιατί δεν είναι και πολύ λογικό αυτό. Η κυρία Καρβάλιο. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρουσιάσεις. Θα ήθελα να κάνω μια υπόδειξη και θα ήθελα τη δική σας γνώμη. Ένας ε, τρόπος για να αυξήσουμε το δίκτυο επιτυχίας, γιατί το 13,8% είναι πολύ χαμηλό, υπάρχουν πολλές ε, καλές προτάσεις, που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί είναι να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας άλλος τρόπος θα ήταν σε εθελούσια βάση τα, οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τις προτάσεις που ήταν ε, επιτυχής ε, μέσα στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων ή άλλων ευρωπαϊκών ταμείων. Βεβαίως θα πρέπει να γίνει σε θελούσια βάση, αλλά αν ε, μερικά κράτη αρχίσουν τότε οι άλλοι θα, τα υπόλοιπα κράτη δεν θα θέλουν να μείνουν πίσω. Και αυτό θα αποτελέσει έναν απλό τρόπο για να φτάσουμε σε έναν κοινό χώρο έρευνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μία αποτίμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη. Έτσι ώστε να υπάρχει υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, αριστεία στην Ευρώπη, όχι μόνο από αυτές τις περιφέρειες αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δηλαδή να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ε, πάνελ το οποίο να συσταθεί με κριτήρια αριστείας έτσι ώστε να υπάρχει και λιγότερη γραφειοκρατία να μην χρειάζεται να δαπανώνται κονδύλια για μια εξεταστική επιτροπή θα μπορούσαν να κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να συνεργαστούν έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε περισσότερα ε, ευρωπαϊκά σχέδια με αυτή τη διαδικασία επιδότησης υποτροφιών. Ματίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις και θα ήθελα να επιμείνω ε, για ένα θέμα που έθιξε η καθηγήτρια Νοβότνη και άλλοι συνάδελφοι σε σχέση με την αύξηση των υποψηφιών και επιτυχία των κρατών που υποεκπροσωπούνται ή περιφερειών που υποεκπροσωπούνται, διότι δεν αποτελεί απλό στόχο αλλά αναγκαιότητα για να υπάρχει μεγαλύτερη σύνοχη σε ένα τέτοιο μεγαλεπίβολο σχέδιο που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι επιτυχές και με απτά αποτελέσματα. Επειδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα είναι αυτόνομο, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες πολιτικές και στρατηγικές θα ορίσετε για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε σε αυτό το στόχο σε σχέση με τα αρνητικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να επιλύσετε. Η κυρία Μαντουρέλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και να τους συγχαρώ για την εργασία τους. Θα ήθελα να υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Ίσως δεν είναι ε, ερωτήσεις, αλλά περισσότερο ανησυχίες. Η κυρία Νοβότη... Κυρία Νοβότη, γνωρίζετε πολύ καλά τον κόσμο της έρευνας και της επιστημονικής κοινότητας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι νομίζετε ότι σκέφτονται οι ερευνητές μας μετά από αυτό το διάστημα λειτουργίας του Συμβουλίου Έρευνας και αν νομίζετε ότι η επιστημονική μας κοινότητα πιστεύει ότι ανταποκρίνεστε στις προσδοκίες γιατί εμείς ε, έχουμε διαφορετικές γνώμες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε στοιχεία από αυτού. Δηλαδή αυτό που με, μας ενδιαφέρει είναι η κοινωνική αποτίμηση. Έχουμε να κάνουμε με μία απτή πραγματικότητα. Είπατε ότι δεν ευεργετήθηκαν όλα τα κράτη-μέλη από τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και αυτό οδηγεί σε αδιαφορία, σε μερική αδιαφορία από τα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει και την λειτουργία του ERC εάν δεν είναι ενθουσιώδης ε, δηλαδή η επιστημονική κοινότητα. Δεν θα πρέπει να εξεύρουμε έναν τρόπο έτσι ώστε να λειτουργήσουμε βάση την αριστεία, αλλά να μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότεροι. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θα πρέπει να καλύψει τα χάσματα που υπάρχουν στον οικονομικό, εδαφικό και κοινωνικό τομέα για να υπάρχει ίση πρόσβαση για όλους. Και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να συντάξουμε όλες ε, τις ε, τεχνολογικές ε, κοινότητες. Ευχαριστώ, κύριε Νοβότνη. θα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Ναι. Ναι, ναι, από αυτό το μικρόφωνο πρέπει να μιλήσω, έτσι μου είπαν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σχολιάσω το ζήτημα που σας απασχόλησε περισσότερο από όλο. Σας διαβεβαιώ ότι και εμείς πιστεύουμε ότι τα καλύτερα επιστημονικά μυαλά και ταλέντα βρίσκονται παντού στην Ευρώπη. Η καθηγήτρια Μουνιέ γεννήθηκε στη Ρουμανία και ένα μέρος της εκπαίδευσής της έγινε εκεί και τώρα εργάζεται στην Γερμανία. Δυστυχώς αυτό ισχύει για πολλούς νέους σε αυτές τις χώρες. Εσείς θα έχετε τους προσωπικούς σας λόγους προφανώς, αλλά ας δούμε κι εμείς κάποιους από αυτούς τους λόγους. Δηλαδή, η σχέση ανάμεσα στις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτών των χωρών, η κατάσταση προς την κατάσταση των πανεπιστημίων, υπάρχει στενή σχέση δηλαδή ανάμεσα στο ύψος των δαπανών μιας χώρας για την έρευνα και την ανάπτυξη ε, και το, ε, σχέση με τον αριθμό των υποτρόφων λοιπόν ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ερεύνας. Εάν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ψηφίζουν με τα πόδια τους, είναι, πηγαίνουν αλλού, τα μαζεύουν και πηγαίνουν αλλού. όποιος ε, απευθύνεται σε μας και μας ε, ε, θέτει αυτό το ερώτημα θα το απαντήσουμε το ίδιο ότι η βασική μας αρχή είναι η αριστεία γιατί αυτός είναι ο στόχος μας θέλουμε να χρηματοδοτούμε εξαιρετικούς ερευνητές για να διεξαγάγουν εξαιρετική έρευνα Άρα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό που βλέπουμε ότι χώρες, ε, και μπορώ να ε, αναφερθώ σε μια μεγάλη χώρα, την Πολωνία, που πρόσφατα ίδρυσε έναν οργανισμό ε, εμπνεόμενη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για να ανεβάζει το επίπεδο στη διαδικασία επιλογής για την Πολωνία ακολουθείται μια πολιτική επιλογής αξιοκρατική, Όπω θα έπρεπε να είναι. Οπότε, μεσοπρόθεσμα, ευελπιστούμε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα καρποφορήσουν και οι νέοι, αν δουν, διαπιστώσουν ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση στις χώρες του, θα έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν. Να το επιθυμούν βέβαια Δεύτερον, θα ήθελα να απαντήσω ε, στην ερώτηση της κυρίας Καρβάλιο. Αυτό γίνεται ήδη μπορώ να σας πω με τα χαράς αλλά σε εθελοντική βάση. Μετά τον πρώτο ε, γύρο των αρχικών υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας είπαν ναι, κάποιες χώρες ότι όσοι είχαν κληθεί για προσωπικές συνεντεύξεις, γιατί έτσι αρχίζουμε για τις αρχικές υποτροφίες, βρίσκονται σε τόσο υψηλό επίπεδο αριστείας ε, που θα τους δεχτούμε έτσι και θα τους χρηματοδοτήσουμε. Βεβαίω, ε, η χρηματοδότηση προέρχεται και από εθνικέ πηγέ, και κάποιε χώρε ε, συνεχίζουν, άλλε πάλι όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση Νομίζω ότι οι χώρες μας θα πρέπει να ε, αποδώσουν τη δέουσα σημασία σε αυτή την πρωτοβουλία διότι είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο και θα ενθαρρύνουν με αυτόν τον τρόπο τους ερευνητές τους. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι για την ανεξαρτησία, την αυτονομία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνα και παρεμπιπτόντω να σα ευχαριστήσω για την προηγούμενη στήριξη που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κατοχυρωθεί και να ενισχυθεί η ανεξαρτησία, η αυτονομία του Συμβουλίου Έρευνας. Ο Ζακ μετά την έκθεση της κυρίας Φρέιμπεργκερ, ε, μετά την εφαρμογή της έκθεσης δηλαδή, μας είπε ότι ε, τις υπόλοιπες εκθέσεις τις εξετάζει η Task Force, η ειδική ομάδα και τα αποτελέσματα αναμένονται για τις πρώτες ε, δύο εβδομάδες του Ιουλίου. Δεν είναι ότι στο παρελθόν δεν υπήρξαν προβλήματα αλλά οι σχέσεις ε, με την εκτελεστική υπηρεσία είναι πλέον αρμονικές και συνεργαζόμαστε για την επίτευξη κοινού στόχου και τα υπολοιπόμενα ε, δομικά προβλήματα θα τα εξετάσει και θα τα ρυθμίσει η Task Force. Κάτι άλλο εδώ που βρίσκω ενδιαφέρον ε, Αυτά που είπατε για την ε, ερευνητική αριστεία και την αριστεία στον τομέα της καινοτομίας. Ε, ποιος κρίνει την αριστεία για την επιστημονική αριστεία είναι πολύ απλή απάντηση. Ε, εκτίμηση, αποτίμηση ομοτήμων, peer review. Οι καλύτεροι δηλαδή επιστήμονες κρίνουν τα προγράμματα, τις ε, προτάσεις βάσει διεθνών προτύπων και για την ε, αριστεία στον τομέα της καινοτομία είναι η ίδια αγορά και η κοινωνία. Γιατί τι σημαίνει καινοτομία, ότι υιοθετείται μία ιδέα, αν πρόκειται για τεχνολογική καινοτομία, υιοθετείται από την αγορά αυτή η ιδέα, πρόκειται για μία διαδικασία ή ένα προϊόν, ένα αγαθό ή αν πρόκειται για καινοτομία κοινωνική, υιοθετεί την ιδέα η ίδια η κοινωνία, το κοινωνικό σώμα. Οπότε αυτοί θα είναι και οι κριτές της αριστείας στον τομέα της καινοτομίας και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να και η κυρία καθηγήτρια. Ναι, σύντομα. Ήθελα να πω πως όταν έφυγα εγώ από τη Ρουμανία ήταν εξαιρετική εκπαίδευση. Πήδηξα δύο τάξεις στη Γερμανία και τελείωσα αμέσως ε, το Λύκειο. Οπότε θα ήθελα να δώσω, να προσφέρω κάτι στον τόπο καταγωγής μου. Πήγα ε, πίσω στη Ρουμανία να στήσω ένα μεταπτυχιακό. Απλά στο εργαστήριό μου έχω 25 άτομα, 18 από τους οποίους είναι από το εξωτερικό, από την Ανατολική Ευρώπη και από την Ιταλία και τη Γαλλία. Το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα και πρέπει να γίνει κάτι στη χώρα για να προσελκύσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν εργαστεί στα καλύτερα ιδρύματα της Δυτικής Ευρώπης, στο εργαστήριό μου, στο Ινστιτούτο Max Planck και Εξεπλάγιν ναι, και όταν επισκέφθηκα πρόσφατα ένα Ινστιτούτο στο Βουδαπέστη και στον δικό μου τον τομέα υπάρχει ένα Ινστιτούτο στη Βουδαπέστη που είναι κορυφαίο πραγματικά, μπορεί να ανταγωνιστεί με οποιοδήποτε διεθνές ε, ίδρυμα και έχουν τους καλύτερους ερευνητές ε, στην Euroscience και μάλιστα έχουν ζητήσει και έχουν λάβει πάρα πολλές επιχορηγήσεις και από το Ευρωπαϊκό η ίδρυμα έρευνας είναι δυνατόν αλλά πρέπει να καταστεί δυνατόν εκεί να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Και η Γερμανία είχε το ίδιο πρόβλημα. Έχανε πάρα πολύ κόσμο που πήγαινε στις ΗΠΑ και είναι τώρα η ευκαιρία να τους έχει πίσω. Και μάλιστα η Γερμανία καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να ενθαρρύνει τον κόσμο να ζητήσει ε, έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο Έρευνας γιατί δεν το κάνουν αρκετά αλλά είναι δυνατόν και πρέπει κάτι να γίνει για να πάνε οι άνθρωποι αυτοί πίσω στις ε, χώρες τους. Οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν. Να προσθέσω εδώ πέρα πως ε, πίσω από κάθε υπότροφο που βλέπετε υπάρχουν 4-5 διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί που προσλαμβάνονται με τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γιατί ένα 70% πηγαίνει σε κόστος μισολογικό, είναι νέοι άνθρωποι διεθνείς στον προσανατολισμό τους, οπότε τα νούμερα τα οποία σας έδωσα τα πολλαπλασιάζετε επί 4, επί 5 και έχετε μια μελλοντική γενεά εξαιρετικά εκπαιδευμένων ερευνητών που συνεργάζονται με τους υποτρόφους μας. Και για να επανέλθω στο ερώτημά σας, νομίζω πως έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία εντός της επιστημονικής κοινότητας και αυτό ταυτόχρονα είναι και το ισχυρό μας σημείο. Έχουμε ρίζες στην επιστημονική κοινότητα, για αυτούς εργαζόμαστε και το εκτιμά αυτό η επιστημονική κοινότητα και ελπίζουμε να προσφέρουμε και στην κοινωνία αυτά τα οποία επενδύει σε μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν και ενδιαφέρουσες και ε, θετικές αυτές οι ειδήσει και νομίζω πως ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να έχουμε κάποιον ο οποίος θα μας πει πόσο υποφελείται από το, συστήματα, από το σύστημα. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες μου, κύριοι και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Και συνεχίζουμε με την έρευνα σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Από τις προκλήσεις της ευκαιρίες προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, η κυρία Ματίας έχει το λόγο. Έχετε το λόγο. If you want. Αν θέλετε. Σας ευχαριστώ. Φυσικά και θέλω το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι όμως σύντομη. Η συζήτησή μας εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων συζητήσεων σήμερα το απόγευμα μέσα στα πλαίσια του κοινού πλαισίου στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Θα ήθελα να σας σκιαγραφίσω τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν το σχέδιο έκθεσης. Όλοι το έχετε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες λοιπόν. Καταρχήν να πω ότι έχει μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση μέσα στα πλαίσια των επόμενων δημοσιονομικών πρόπτικων για να ορίσουμε το κατάλληλο πλαίσιο χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Δεύτερον, να πω ότι κατανοώ ότι η έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία μας απασχολούν ως προς την προτινόμενη, προστιθέμενη αξία και αυτό που έχει σημασία είναι ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε αναγνωρίζοντας αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και εδώ υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές. Άρα, με βάση τις προτάσεις της πράσινης βίβλου, προβλέπω μία επανοργάνωση του συστήματος. Έχουμε μέσα τρόπους χρηματοδότησης, συμμετέχοντες. Θα πρέπει να καλύψουμε ορισμένα από τα χάσματα που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θα πρέπει να ορίσουμε εκ νέου αυτή τη στρατηγική, να την τελειοποιήσουμε. Θα πρέπει να την εκλάβουμε ως μια ευκαιρία με βάση τα όσα συζητήθηκαν εδώ ως προς την απλούστευση της έρευνας, την ενδιάμεση αξιολόγηση μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου και η αποτίμηση της καινοτομίας. Έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία θα ενισχυθεί. Άρα με βάση αυτά που μας παρουσίασε η Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο και με βάση τα τρία προγράμματα, πρόγραμμα πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας καθώς και με τα διαρθρωτικά ε, ταμεία και με το Ταμείο Συνοχής για την έρευνα και την καινοτομία, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επανοργωνώσουμε αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο χρηματοδότησης. Θα πρέπει να ξέρουμε να επιμερίζουμε για να φτάνουμε σε ένα κοινό σύνολο και να αξιολογήσουμε καλύτερα τους, αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας θα πρέπει να δεχόμαστε το διαφορετικό. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως ισότιμο ή ίσο αυτό που είναι διαφορετικό. Δηλαδή ως προς τα πανεπιστήμια ή τις ΜΜΕ ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να τα εξομοιώνουμε όλα αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά για να αξιολογήσουμε και την προστιθέμενη αξία της έρευνας και της καινοτομίας. Μετά από όλα αυτά, πιστεύω ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε ορισμένα ζητήματα. Βρισκόμαστε στην απαρχή της συζήτησης. Αυτό το προσχέδιο ορίζει κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες θα εμβαθύνουμε. Υπάρχουν όμως ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Η πράσινη βίβλος βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, στην αριστεία, στα αποτελέσματα. Άρα όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, αριστεία και έρευνα θα πρέπει να γνωρίζουμε κατά πόσο προωθούμε πραγματικά την αριστεία ή τους άριστους που υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το ίδιο αφορά τα αποτελέσματα. Εάν βασιζόμαστε στα αποτελέσματα της έρευνας, θα πρέπει να είμαστε σαφείς, γιατί πολλές φορές ο ερευνητής την χάνει αναγνώρισης, έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις, προωθεί ένα αγαθό ή ένα εμπόρευμα. Άρα δεν πρέπει να ε, κρίνουμε ως ίσο ή η ισότιμο αυτό που είναι διαφορετικό. Υπάρχουν πιο ολοκληρωμένες οικονομίες και περιφερειακές οικονομίες. Άρα το σχέδιο ευρωπαϊκής σύγκλησης έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ε, μέσα στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων μπορούμε να προωθήσουμε συγκεκριμένα έργα. Δηλαδή είμαστε υπέρ της αριστείας αλλά όχι κατά της σύγκλησης και της συνοχής Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον συγκεντρωτισμό πόρων και μέσων. Μιλήσαμε για ένα 50% των υποτροφιών που χορηγούνται μόνο σε 40 Ινστιτούτα. Αυτό κάτι σημαίνει στα πλαίσια της Ευρώπης που ζούμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την συμμετοχή των κρατών μελών και των περιφερειών που υποεκπροσωπούνται. Και αυτό αφορά τα νέα κράτη-μέλη και τις χώρες του Νότου. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής ανάλογα με τον ε, τύπο των συμμετοχών και των συμμετεχόντων. Θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες και όχι να δημιουργούνται προσκόμματα. Αυτά είναι τα γενικά στοιχεία. Για τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουμε. Θα πρέπει να αρκεστούμε σε τρία επίπεδα. Λοιπόν, να δούμε τι είναι πραγματικά, να διαχωρίσουμε την έρευνα από την καινοτομία και μέσα στην καινοτομία να δούμε ποια είναι η καινοτομία, η κοινωνική ε, καινοτομία και ποια στρέφεται προς την αγορά. Επίσης, να αυξήσουμε τις ικανότητές μας και να επαυξήσουμε τις υποδομές. Θα πρέπει να προωθήσουμε σχέδια ευρείας κλίμακας, να υπάρχουν ειδικέ γραμμές στον προπολογισμό όπως για τον Γαλιλαίο Ίτερ και άλλα που θα πρέπει να βγουν από το πρόγραμμα πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας, Ανάπτυξης και Τεχνολογίας θα πρέπει να λαμβάνει και επιδοτήσεις από την ΕΤΕ και χρηματοδότηση από την ΕΤΕ. Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης δανειοδότησης και ως προς τα ειδικά προγράμματα ικανοτήτων θα πρέπει να προωθήσουμε και τις πρωτοβουλίες Marie Curie. σε συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία. Ένα δεύτερο επίπεδο αφορά την παγιοποίηση αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο για την αξιοποίηση της έρευνας. Θα πρέπει να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας και δυνατότητες για να προωθήσουμε την ε, ε, έρευνα σε διαπανεπιστημιακό επίπεδο και θα πρέπει να έχουμε χώρο για τους διάφορους τομείς, να υπάρχει μια διατομιακή δηλαδή έρευνα. Να ε, διπλασιάσουμε δηλαδή τον προϋπολογισμό για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο και με τη χορήγηση υποτροφιών. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, το πρόγραμμα Marie Curie, καθώς και την εργασία των ερευνητών θα πρέπει να εγγυηθούμε μεγαλύτερη σύγκληση και καλύτερη συμμετοχή των γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική διάσταση που πολλές φορές ξεχνάμε. Ένα τρίτο επίπεδο στα πλαίσια αυτής της τροματοποίησης αφορά την καινοτομία και την αγορά. Αυτό τον προσανατολισμό θα πρέπει να προωθήσουμε τις ΜΜΕ που προβάλλουν καινοτομίες. Δυστυχώς υπάρχει χαμηλή συμμετοχή των ΜΜΕ διότι δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα μέσα για να έχουν μια πιο ουσιαστική συμμετοχή. Γι' αυτό προτείνω ένα νέο μέσο χρηματοδότησης για, τα, για τις ΜΜΕ, μία ΕΤΕ δηλαδή, με συγκεκριμένα σχέδια δανειοδότησης που να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ΜΜΕ που προσωπούν την μίζωνα πλειοψηφία, τη συντριπτική ε, πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να τις προσελκύσουμε, γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι αυτή η διάσταση δεν ε, την χάνει, μάλλον αυτή η δεν υπάρχει καν τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει σωστή εκπροσώπηση των ΜΜΕ. Επίσης, η καινοτομία δεν προκύπτει πάντα από την έρευνα. Και κάθε έρευνα δεν οδηγεί σε καινοτομία ή εμπορικά αγαθά. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα κεκτημένα στον ευρωπαϊκό χώρο, ποια είναι τα δημόσια αγαθά που μπορούμε να προωθήσουμε, έτσι ώστε να προωθήσουμε αγαθά, εμπορεύματα και ε, υπηρεσίες που να μπορούν να μπουν στην αγορά. Γι' αυτό Θα ήθελα και τις δικές σας υποδείξεις γιατί υπάρχει πολλής ε, δρόμος μπροστά μας. Ελπίζω να ανακύψει μια κοινή πρόταση του Κοινοβουλίου και να συνεχίσουμε με βάση τις προγενέστερες θέσεις μας στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στη συζήτηση να καλωσορίσω κάποιον τον Γενικό Διευθυντή Αυτοπροσώπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που επιδεικνύεται τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα ζητήματα και είστε εδώ κάθε φορά. Να δώσω τον λόγο λοιπόν στον κύριο Έλερ. Εγώ δεν θα ήθελα να ξεκινήσω με τις συνήθεις ευχαριστίες, αλλά ε, τις συνήθεις τυπικές ευχαριστίες, αλλά να ευχαριστήσω στα αλήθεια την εισηγήτρια. Γιατί θεωρώ πως παρά τις ιδεολογικές διαφορές ε, ε, μεταξύ εισηγήτριας και ημών των σκιωδών είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και υποβάλαμε μια έξυπνη και θαραλέα, ένα έξυπνο και θαραλέο σχέδιο έκθεσης. Να κάνω κάποιες συμπληρωματικές λοιπόν παρατηρήσεις. Πρώτον, ποιο μπορεί να είναι το μήνυμα της πράσινης βίβλου. Η πράσινη βίβλος θα είναι στην αγορά, αν θέλετε, θα βγει στην αγορά, στο μέσο της ε, πολιετούς ε, συμφωνίας, των διαπραγματεύσεων της πολιετούς συμφωνίας και βεβαίω αυτός είναι ο ρόλος του και είναι σημαντικό να επαναλάβουμε και προς την Κομισιόν και προς το Συμβούλιο πως συμφωνούμε πως ε, και στην Πράσινη Βίβλο υπάρχει η αίτηση να διπλασιάσουμε τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεύτερον είναι ένα από τα κεντρικά σημεία που επεξεργαστήκαμε μαζί με την κυρία Καρδάγιο, ότι δηλαδή επαναλαμβάνουμε πως πριν μπούμε στην ουσία ενός άλλου προγράμματος πλαισίου, συμφωνούμε πως η απλοποίηση είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα πριν μιλήσουμε για επανασχεδιασμό προγράμματος πλαισίου. Τρίτον, θεωρώ πως είναι σημαντικό όταν συζητάμε ζητήματα όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μιλήσουμε πραγματικά για κάποια κατά συνθήκη ψεύδη που επικρατούν σε αυτό το τομέα. Δηλαδή με υπάρχοντα ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εάν μιλάμε συγκεκριμένα για τομείς θα οδηγήσει το πρόγραμμα αυτό στη μη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί κάπου έχουμε ε, επιλέξει ορισμό που είναι πάρα πολύ μικρός, πολύ χαμηλός και ε, από την άλλη υπάρχουν κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις με μεγάλη καινοτομία οι οποίες αποκλείονται από την άλλη θεωρώ πως ε, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να βρούμε μια λύση. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο δεν αναφέρεται στην έκθεση. Είναι το Risk Sharing Facility. Το Κοινοβούλιο έχει μια, υποστήριξε μια πειραματική προσέγγιση αλλά βεβαίως όσον αφορά αυτό δεν θα δίνουμε μόνο τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις, τις μεγάλες βιομηχανίες, αλλά θέλουμε το Risk Sharing Facility να χρησιμοποιείται διαφορετικά, να υπάρχουν και εθνική ενδιάμεση, να είναι γνωστό πως ε, υπάρχει μια διαφορετική χρηματοδότηση, να μην υπάρχει η ψευδέστηση πως είναι κάτι το οποίο θα στηρίξει γενικά την οικονομία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε να τονίσω μια τελευταία πτυχή. Με την Κομισιόν πιστεύω συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά να το ξεκαθαρίσω. Η πορεία αυτή ορίζεται ως εξής, σε αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν με την Πράσινη Βίβλο και γνωρίζουμε πως στο εσωτερικό της Κομισιόν υπάρχουν πολύ πιο προχωρημένες σκέψεις ως προς το θέμα αυτό. Ίσως οι δύο σημαντικότερες ε, προσεγγίσεις είναι αφενός το θέμα της καινοτομίας. Θεωρώ πως εδώ πέρα μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά με έναν σαφή ορισμό του που οδηγεί αυτό το πράγμα. Γιατί αν έχουμε πάλι κάτι το αφηρημένο, δεν είμαστε διατεθειμένοι π.χ. να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ε, μια πρώτο καθεδρία στην επιστημονική αριστεία. Τι σημαίνει η επιστημονική αριστεία γιατί σημαίνει επίσης αριστεία στην ε, καινοτομία. Επίσης το ίδιο ε, για την συνένωση προγραμμάτων σε ένα κοινό μεγάλο πρόγραμμα. Οπότε απαιτούνται δραστικά ε, βήματα μεταξύ του προγράμματος πλαισίου 7 και 8, αλλά πρέπει να είναι σαφές πως δεν θα υποστηρίζαμε ε, κάτι το οποίο θα αμφισβητούσε παραδείγματος χάρη την ε, ομαδική ε, έρευνα. Αυτό αν αμφισβητηθεί νομίζω κάτι τέτοιο είναι πολύ σοβαρό όπως και το ζήτημα των προγραμμάτων συνεργασίας. Οπότε νομίζω πως έτσι όπως έχουν τα πράγματα έχουμε μια πάρα πολύ καλή πρώτα, ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο έκθεσης και πρέπει να επικεντρωθούμε στο να στείλουμε τα σημαντικά μηνύματα το Σεπτέμβριο και θα έχουμε βέβαια δυνατότητα να έχουμε κάποια διαφοροποίηση αλλά θεωρώ πως είναι σημαντικό το να έχει κοινή θέση το Κοινοβούλιο γιατί μπήκαμε κάπως αργά στη διαδικασία του προγράμματος πλαισίου 7 και όσον αφορά την Πράσινη Βίβλα τουλάχιστον ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο τέλος από πλευράς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος μαζί με τους συναδέλφους τους σοσιαλδημοκράτες ε, εισάγαμε εδώ πέρα για πρώτη φορά μία έννοια ονόματι Stairway to Excellence. Δηλαδή βλέπουμε πώς ακριβώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν και οι νέες χώρες. Και εδώ πέρα ακριβώς εφαρμόζονται δύο πράγματα. Αφενός το ότι θέλουμε να μείνουμε στην αριστεία, αλλά και να αναζητήσουμε τρόπους συμμετοχής ε, και ενίσχυσης των νέων χωρών. Όμως ο συμβασμός σημαίνει πως δίνουμε βάρος στην αριστεία, γιατί οτιδήποτε άλλο θα αμφισβητήσει τις αρχές του προγράμματος και είναι σημαντικός ο συμβιβασμός γιατί πρέπει να προσέξουμε το θέμα είναι να ενισχύσουμε την καινοτομία στις νέες χώρες, αλλά όχι να γίνει το πρόγραμμα αυτό πρόγραμμα συνοχής. Το επαναλαμβάνω αυτό. Είναι κεντρικός πυλώνας της πολιτικής μας στάσης. Δεν μπορούμε όλα τα προγράμματα της Ευρώπης να γίνουν προγράμματα συνοχής. Πρέπει η Ευρώπη να είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Και όταν μιλάμε για διεθνή ανταγωνισμό δεν ασχολείται κανείς με τη συνοχή, ανταγωνιζόμαστε με την Ασία και τη Βόρειο Αμερική. Με το Stairway to Excellence όμως δεν έχουμε βρει μόνο μια ωραία λέξη, αλλά θέλουμε να κάνουμε και κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και όχι μόνο για τους παλαιούς 15 αλλά και για τις 27 χώρες και πρέπει βεβαίως να στείλουμε ένα μήνυμα υπέρ της καινοτομίας και της έρευνας στην Ευρώπη με την αύξηση των κονδυλίων για το πρόγραμμα πλαίσιο 8. Η κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας. Έχετε ε, προβάλει ε, ιδιαίτερα σημεία ως προς την έρευνα και την καινοτομία για να υποστηρίξω αυτά που ελέγχθησαν. Είμαι πολύ απογοητευμένη διότι όλη μας η εργασία για την έκθεση Καρβάλιο που υπήρχε μεγάλη ομοφωνία από το Κοινοβούλιο όλη αυτή η εργασία δεν ελήφθη υπόψη από την Κομισιόν. Ελπίζω λοιπόν η εργασία μας εδώ να ληφθεί υπόψη από την Κομισιόν γιατί πολύ σπάνια είναι ομόφωνο το κοινοβούλιο για μια έκθεση. Πολλοί χτυπούν ε, και το λάθος κουμπί, ακόμα και όταν θέλουν να είναι ομόφωνοι. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα σωστά κονδύλια πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση από τους ερευνητές, τους επιστήμονες που δουλεύουν σε εργαστήρια, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν προς λάθος, τη λάθος κατεύθυνση αυτά τα κονδύλια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε. Έχουμε ένα στόχο Στόχος μας δεν είναι να αυξήσουμε τις δαπάνες στο 3% για την έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε να αυξήσουμε τα κονδύλια για την έρευνα και την ανάπτυξη για να ε, έχουμε ε, τεχνολογίες εχμής, να προωθήσουμε τους δείκτες ανάπτυξης και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια υπέρ της έρευνας και ανάπτυξης. Και νομίζω όταν μιλώ σε επιστήμονες και ερευνητές βλέπω ότι υπάρχει μία συνεργατική στάση και με την βιομηχανία, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, φιλανθρωπικές οργανώσεις κλπ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε ο φορολογούμενος να μην καταβάλει άδικα τα χρήματα και να εργάζεται ε, περισσότερο με τη θέλησή του. Μιλήσαμε για ΜΜΕ πράγματι, θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι, ότι δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, ε, γιατί όταν πάνε τα κονδυλία στις μεγάλες επιχειρήσεις ε, μπορείτε να το αιτιολογήσετε αιτιολογήσετε αλλά δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε για λάθος λόγους τις επενδύσεις και ορισμένες φορές αυτό που γίνεται ιδιαίτερα αρεστό από αυτά τα προγράμματα είναι ακριβώς αυτή η διάσταση ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αριστεία, μάλιστα. Ε, πιστεύω ότι οι παρουσιάσεις παρου... Ε, πραγματεύτηκαν σωστά το ζήτημα και φυσικά θέλουμε να εκπληρώσουμε το στόχο της καινοτομία, αλλά να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις. Αυτή η ιδέα σχετικά με το stairway, με την ε, σκάλα προς την αριστεία, ναι θετικά όλα αυτά, να ενθαρρύνουμε τους νέους από διάφορες χώρες, να βοηθήσουμε τις λεγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, αλλά το σημαντικό εδώ είναι η σχέση με το Ταμείο συνοχή ε, και με την δομή του οργανισμού. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια ε, ε, πλουσίων χωρών που διοχετεύουν περισσότερα κονδύλια ε, στα προγράμματα και ε, ούτως ή άλλως δεν λαμβάνουν τα ίδια ποσά από άλλες χώρες από το Ταμείο Συνοχής. Ε, γίνεται μια αντιστάθμιση. Δηλαδή πάντως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να λειτουργεί η χρηματοδότηση πιο αποτελεσματικά. Βεβαίως τώρα ζούμε την κρίση και χρειάζεται να λειτουργούμε πιο έξυπνα και να συνδυάζουμε πιο έξυπνο τρόπο τα διάφορα Αρθρωτικά ταμεία, μιλήσατε για τα soft loans, μιλήσατε για τις ε, ε, χορηγίες. Με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρύνουμε τις επιχειρήσεις. Um, sorry, maybe slightly, slightly jumping, jumping around your report. Uh, από το ένα στο άλλο, αλλά τέλος πάντων θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους νέους ερευνητές. Ε, αλλά πέρα από αυτό, ε, όλοι περιμένουν να κάτσουμε να δουλεύουμε μέχρι με μεγάλης ηλικίας ε, αλλά ήθελα, το λέω αυτό γιατί πρέπει να προσέξουμε τη διατύπωση. Δηλαδή μην να τους αποθαρρύνουμε τους πιο ηλικιωμένους γιατί είναι σοφοί. Μην το παραγνωρίζουμε τη σημασία αυτού και να εστιάζουμε μόνο στους νέους. Ένα λεπτό και τώρα απευθύνομαι και στην Επιτροπή γιατί ξέρω ότι με ακούνε. Ε, προς το τέλος της έκθεσης υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες παράγραφοι, 25 παραδείγματος χάρη, λέει ότι δεν έχουμε ενισχύσει τον ανταγωνισμό παρότι έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, με το πρόγραμμα συνεργασίας μέχρι το 2025. Ε, στην ε, παράγραφο 27 έχουμε τα προγράμματα που ξεκινάνε από κάτω προς τα πάνω και τα άλλα που ξεκινάνε από πάνω προς τα κάτω. And, Και στην παράγραφο 28 απευθύνουμε την έκκληση για διεθνή συνεργασία όπου δει, λέμε. Πρέπει να προσθέσουμε ότι πρέπει να γίνεται μόνο όταν χρειάζεται. Η διεθνή συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε αριστεία, σε εξαιρετικέ ιδέε, αλλά όχι σε όλε τι περιπτώσει. Ε, θα ήθελα να υποβάλω τροπολογίε για το, την παράγραφο σχετικά με το άρθρο 15. Τι θέλουμε να κάνουμε με τις σταδιοδρομίες των ερευνητών. Μιλήσατε για επισφαλή κατάσταση για τους ερευνητές, αλλά δύσκολα εγώ μπορώ να έχω μια εικόνα του τι εννοούμε. Ξέρετε τι εννοούμε. Εννοούμε ότι διερευνούμε για ποιο λόγο ε, μπαίνουν στον πειρασμό να φύγουν από την Ευρώπη οι ερευνητές. Γιατί αυτό συμβαίνει. Οι ε, καλύτεροι ερευνητές πάνε στη ΣΥΠΑ, πάνε στην Κίνα. Πρέπει να δούμε λοιπόν για ποιο λόγο. οι ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία που χρειάζονται. αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Πρόκειται για επισφαλή θέση εργασία. Μην χρησιμοποιούμε του ίδιου όρου. Αυτό το precarious workers που είπατε. Ε, ε, ε, δεν αρμόζει γιατί ο άλλος είναι ο στόχος μας. Εμείς θέλουμε να παραμείνουν στις θέσεις τους οι ερευνητές. Αυτά και περιμένω τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ κυρία Ριέρα Μαντουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ματίας. Ευχαριστώ για την δουλειά σας και τις εξηγήσεις σας. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις, ε, να προσθέσω κάποια σχόλια σε αυτά τα οποία μας είπε η κυρία Ματίας. Γενικά συμφωνώ με αυτά τα οποία ακούστηκαν ήδη. αναφερθώ στην χρηματοδότηση για ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο ε, χρηματοδότησης ε, που πρέπει να αποφασίσουμε ε, το ότι πρέπει να διατηρήσουμε το κοινωνικό μας μοντέλο. Για να γίνει αυτό πρέπει να αυξήσουμε τα κονδύλια τι δίνουμε στην έρευνα και να βρούμε νέα λεφτά. Δεν μιλάω για να αλλάζουμε λεφτά, να το πάμε από το νέο τύλο στον άλλον νομίζω πως θα πρέπει να ορίσουμε ξεκάθαρα λεφτά στον προϋπολογισμό μας για αυτές τις πολιτικές και μόνο εάν γίνει κάτι τέτοιο μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Νομίζω πως η κυρία Ματίας μας τα είπε σωστά και νομίζω πως είναι κάτι που μπορούν να στηρίξουν όλες οι ομάδες στην Επιτροπή μας. Επίσης, ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τη δομή που θα θέλαμε στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Να είμαι σαφής. Νομίζω πως ένα πρόγραμμα πλαίσιο το οποίο έχει μια πιο διεπιστημονική δομή θα πρέπει να είναι δυνατόν να λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω. Οι ίδιοι επιστήμονες θα πρέπει να μπορούν να προτείνουν ποια ζητήματα θένε να δούνε. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμετοχή επίσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο δεν έχει επιληθεί. Νομίζω λοιπόν πως πολλά έχουν να, γίνει, έχουν να γίνουν για το να βρούμε και να δοκιμάζουμε νέες ιδέες επίσης όπως είπαν και άλλοι. Θα πρέπει να έχουμε κίνητρα για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου διασυνοριακά με περαιτέρω συνεισφορές από ευρωπαϊκά ταμεία και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη διαφάνεια να υπάρχουν περιορισμένοι κοινοί κανόνες και λιγότερο δυσκίνητες ε, διαδικασίες όσον αφορά δε τα προγράμματα συνεργασίας πρέπει να ενισχυθούν αλλά επίσης πρέπει να δώσουμε βάρος στην βασική έρευνα χωρίς να προσδιορίσουμε συγκεκριμένα σε σχέση δε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λαμβάνουν χρηματοδότηση οι επιστήμονες από όλα τα κράτη-μέλη. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας. Το έχουμε πει αυτό όσον αφορά την κινητικότητα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την κινητικότητα, ειδικά όσον αφορά την βιομηχανία. Πρέπει να ενισχύσουμε τη χρήση διαρθρωτικών κονδυλίων και αυτό για ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα και την βιομηχανία και την διεθνή συνεργασία. Και για να καταλήξω με τα αρχικά μου αυτά σχόλια, θα θέλαμε το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο να συμπεριλαμβάνει και την ε, κοινωνική διάσταση. Είναι κάτι που το φύγουμε συνεχώς και πρέπει να αναπτυχθεί ως οριζόντιο θέμα. Θα σταματήσω εδώ πέρα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Καρβάλιο. Ε, Ευχαριστώ. Και ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Μαρίζα Ματίας. Πολύ καλή έκθεσή της. Τα περισσότερα τα είπαν ήδη οι συνάδελφοι, ο κύριος Έλερ και άλλοι. Θέλω να προσθέσω μόνο τρεις παρατηρήσεις. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η δομή ε, που μας παρουσίασε η Μαρίσα με τα, τις διάφορα, με τα διάφορα στρώματα, ότι δηλαδή θα πρέπει να βρίσκεται το ε, Ινστιτούτο όχι στο πρώτο αλλά στο δεύτερο στρώμα. Δεύτερον, ε, διπλασιασμός των κονδυλίων. και θέλω να αναφερθώ σε κάτι που υπήρχε στην έκθεση της ΣΟΥΡΕ. Ήταν σε μία από τις συμβαστικές ε, τροπολογίες που ελπίζω να υπερψηφίστηκαν σήμερα ε, να ζητήσουμε για ισχυρότερη ε, διακυβέρνηση, καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων. Έχουμε τώρα ισχυρότερη οικονομική διακυβέρνηση. Θα πρέπει να μελετήσουμε το μοντέλο για να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τη χρηματοδότηση της έρευνας. Ούτως ώστε ε, να επομιστούν ε, το δικό τους το κομμάτι τα κράτη-μέλη ως προς τη χρηματοδότηση και να δημιουργηθεί το πλαίσιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας. Είπαμε πολλά για τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στον τομέα της ε, έρευνας για τις υποδομές, τις τεχνολογικές υποδομές. Προφανώς αυτό είναι συνάρτηση των προτεραιοτήτων κάθε κράτους μέλους, αλλά πάντως θα ήταν θετικό να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση στον τομέα της έρευνας ε, στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε μελλοντικά αυτό το ζήτημα γιατί έχει αναφερθεί ε, στην έκθεση Γκαλέκα ε, Γκαρίντα, στην έκθεση δηλαδή της Επιτροπής ΣΟΥΡ. Ευχαριστώ τη Μαρίσα Ματίας για αυτά που είπε για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, για την ε, απλοποίηση. Δεν υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες με στην έκθεση λόγω του περιορισμού του μεγέθους της έκθεσης. Και θα υποβάλω τροπολογίες για αυτό το θέμα, για όσα σημεία ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα στις τροπολογίες μας πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απλούστευση δεν σημαίνει ότι θα έχουμε ίδια μεταχείριση για Ινστιτούτα που διαφέρουν πάρα πολύ, θα έχουμε την ίδια μεταχείριση για ερευνητικά κέντρα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους και ευχαριστώ. Μέρκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Ματίας για τη φιλόδοξη πρώτη παρουσίαση του εγγράφου. Ε, αναγνωρίζω πάρα πολλά πράγματα από την έκθεση περί ένωσης καινοτομίας και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Παρατηρώ πως ε, η, η Επιτροπή να έχει ευθετήσει πολλές από τις ιδέες τις οποίες αναπτύξαμε και την ευχαριστώ. Αναφέρομαι π.χ. στην υπηρεσία μία τάσης για την απλοποίηση των προγραμμάτων και συμφωνώ με τους συναδέλφους πως η απλοποίηση και το να μην υπάρχει τόσος κατακαιρματισμός είναι σημαντικό για τα προγράμματα έρευνας. Πρέπει να γίνουν τα πράγματα πιο απλά με το One Stop Shop λοιπόν το οποίο έχετε πάρει από εμάς σας δίνω συγχαρητήρια επίσης το ότι αναφέρετε την καινοτομία όχι γενικά αλλά ότι υπάρχει τεχνολογική και κοινωνική και ότι έχει και άλλες διαστάσεις σημαντική προσπάθεια γίνεται για ενσωμάτωση της πολιτικής, ε, της ερευνητικής, των διαρθρωτικών ταμείων και των λοιπόν ε, προγραμμάτων. Και υπάρχει σαφής προσανατολισμός το να έχουμε αποτελέσματα στις κοινωνικές ε, προκλήσεις και επίσης για το ότι η Κομισιόν έγραψε κάτι το οποίο μου είναι ιδιαίτερα αγαπητό, δηλαδή την εμπλοκή των πολιτών γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε διάφορα, αλλά εάν αυτά τα πράγματα δεν φτάσουν στην αγορά και στους πολίτες, δεν έχουμε επιτύχει στον στόχο μας, δηλαδή την καινοτομία και δεν θα έχουμε συνεισφέρει. Κατόπιν η φιλοδοξία διπλασιασμού του προϋπολογισμού είναι κάτι το επενετό και να προσθέσω, εντάξει, εμείς μπορεί να τα λέμε αυτά, αλλά όλοι γνωρίζουν πως... Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα, οπότε υποστηρίζω πράγματι το να ζητήσουμε περισσότερα λεφτά για την καινοτομία, αλλά τι θα γίνει όταν θα χρειαστεί να κάνουμε επιλογές, όταν δεν θα μας δώσουν αυτό το προπολογισμό τι, όταν θα πρέπει να διαλέξουμε τι θα στηρίξουμε και τι όχι. Αυτό θέλω να το συζητήσουμε και ίσως μπορεί η συγγήτρια να μας πει λίγα λόγια. Και να δούμε και από πού θα τα βρούμε τα, τα λεφτά για να μείνει ουδέτερος ο προϋπολογισμός σε αυτή την περίπτωση βεβαίως δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα κατόπιν. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο είπε η Μαρίζα Ματίας να υπάρχει δηλαδή μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη και να έχουμε περισσότερη ανοχή όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου που είναι απαραίτητος για την καινοτομία. Και πράγματι να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ μικρών έργων bottom-up και top-down γιατί εδώ πέρα συμφωνώ με τους συναδέλφους πως θα πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές νέες επιχειρήσεις και χρειάζεται να υπάρξει και μια διαφοροποίηση της πολιτικής. Δεν είναι κάθε μικρή επιχείρηση και νέα. Ε, έχουν διαφορετική ε, ομάδα αίματος, αν θέλετε. Even wat, wat punten waar ik wat... Τέλος, κάτι άλλο, ζητήσαμε από την Κομισιόν να ε, φέρει περισσότερα λεφτά στο Risk self Finance Facility και ζητήσαμε από το 1 δισεκατομμύριο να πάμε στα 5. Είναι σαφές πως θέλουμε μεγαλύτερο κομμάτι να πάει σε ένα κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Πώς το βλέπει αυτή την πρόταση η ε, εισηγήτρια, γιατί έχουμε έρευνα και καινοτομία και βλέπουμε πως δεν είναι απολύτως το ίδιο και απαραίτητο το ίδιο αυτά τα δύο πράγματα. Και αναμένω βεβαίως τις επόμενες ε, συζητήσεις και πρέπει πως να πούμε πως η καινοτομία είναι και χρειάζεται διαφορετική πολιτική από την έρευνα, αλλά χρειάζονται και οι δύο. Ευχαριστώ. Έλερ. Er, να προσθέσω κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Στην πράσινη βίβλο είχαμε την κοινή άποψη πως τα μεγάλα ευρωπαϊκά έργα πρέπει να φύγουν από το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Γιατί, γιατί στο έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ήμασταν διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό γνωρίζοντας πως στην φάση της οικοδόμησης δεν θα μπορούσαμε να τα χρηματοδοτήσουμε από το πρόγραμμα αυτό και το ότι υπάρχει διαφορετική γραμμή του προπολογισμού για τα μεγάλα ερευνητικά πρόγραμματα Galileo, GMS e και ITER και το υπόλοιπο ερευνητικό πρόγραμμα είναι κάτι το αποφασιστικό. Αλλιώς δεν θα είμαστε σε θέση τα επόμενα έτη να τρέξουμε αυτά τα προγράμματα και θα έχουμε για το ίτερ, ξέρω εγώ, στο τέλος του χρόνου 700 εκατομμύρια για το GMS, για το Γαλιλαίο τεράστια ποσά. Και τότε το Κοινοβούλιο ήταν έτοιμο για συμβιβασμό την νύχτα του τριμερούς διαλόγου γιατί εμείς δεν θέλαμε να τα σκοτώσουμε αλλά η πραγματικότητα ήταν πως είτε δεν θα υπάρχουν στο μέλλον αυτά τα έργα, είτε θα έχουμε διαφορετική γραμμή του προπολογισμού. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται έτσι. Να δώσω τον λόγο και στο Γενικό Διευθυντή που ακούει τόσο υπομονετικά εκεί πέρα. Good afternoon. Let me first of all... Uh, θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια την κυρία Ματίας. Εξαιρετικό το πρώτο σχέδιο έκθεσης που συντάξατε. Είναι σαφές, ε, είναι ουσιαστικό και βασίζεται και στους ελέγχους για το, την αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο. Αυτά που είπε και η κυρία Καρβάλιο αναφέρεται στην Ένωση για την Καινοτομία και αυτό που έλεγε ο Φανής Τηλερό για πολλά χρόνια, ότι δηλαδή πρέπει να συνδυάσουμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με τα διαρθρωτικά ταμεία. Θα ήθελα να τονίσω την σημασία, όπως και εσείς, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ιδέα αυτή της σκάλας προς την αριστεία Ε, αναφέρετε διάφορα στοιχεία μέσα στην έκθεσή σας ε, για βασικά ζητήματα, για τη δομή τώρα, αυτά, αυτούς τρεις πυλώνες που μας προτείνετε. Ε, είδατε ότι στην πράσινη βιβλό διαφέρει κατά τη δομή που εμείς προτείναμε, αλλά δεν σημαίνει ότι η δική, σας δομή, η δική μας η δομή είναι καλύτερη. Ε, αναφέρεστε στον πρώτο πυλώνα και λέτε ότι είναι ανάπτυξη ε, ενδογενών ε, ικανοτήτων. Ε, capacity building λέτε στα αγγλικά, αλλά αυτό χρησιμοποιείται και στα διαρθρωτικά ταμεία. Οπότε, όπως είπε και ο κύριος Έλερε, θα πρέπει να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Ε, ε δεν μπορούμε να συγχαίουμε δε, τη συνοχή για τα διαρθρωτικά ταμεία με το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε τον τίτλο του πρώτου πυλώνα για να εξασφαλίσουμε με τη συμπληρωματικότητα των διαφόρων μέσων και των πολιτικών, αλλά χωρίς επικαλύψεις. Στην πράσινη βίβλο Αναφερόμαστε εκτεταμένα στους ε, τρεις πυλώνες. Ε, ο ένας βασίζεται στην έρευνα ε, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Ο δεύτερος αναφέρεται στις πολιτικές προκλήσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, για την αποτελεσματική χρήση των πόρων, λύσεις που μπορούμε να βρούμε. Και ο τρίτος πυλώνας είναι ανταγωνιστικότητα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς την ε, ε, ολοκλήρωση του ΣΥΠ τώρα. Είναι λίγο αμφίσιμη η δήλωσή σας, ε, γιατί λέτε ότι είναι προς εξέταση όμως σε προηγούμενες εκθέσεις. Υπάρχουν σαφείς δηλώσεις ότι πρέπει να συνδέσουμε δηλαδή σαφέστατα την έρευνα και την καινοτομία, οπότε είναι σημαντικό το κοινό πλαίσιο να ενσωματώσει το πρόγραμμα πλαίσιο, το πρόγραμμα για την καινοτομία και την έρευνα και το πρόγραμμα για τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική είναι σαφέ ε, ότι αυτό ισχύει και άρα θα πρέπει να κάνει αυτή τη δήλωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορούν ε, να κυκλοφορήσουν στην αγορά τα προϊόντα τη έρευνα και σα είπα βάση των εκθέσεων που ήδη έχουν εγκριθεί. Για τον προπολογισμό δεν χρειάζεται να σα πω, αλλά πολύ ευχάριστο αυτό που λέτε για διπλασιασμό. Τέλο πάντων δεν είναι μέρα τώρα, ούτε ώρα να συζητήσουμε τα κονδύλια. Θα ήθελα μόνο να σχολιάσω τι παρατηρήσει των συναδέλφων σα. Ο κύριο Σέλερ τονίζει πόσο σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι ο βασικό στόχο των διαρθρωτικών ταμείων κατά τη διαστολή με το πρόγραμμα για την καινοτομία, ε, για να αποφύγουμε τι επικαλύψει. Συμφωνώ απολύτω. Επίση είναι σημαντικό τα μεγάλα ε, προγράμματα ε, όπω τον Galileo, το ΙΤΕΡ κτλ., να χρηματοδοτούνται από διαφορετική γραμμή του προπολογισμού και όχι να ανήκουν στο μελλοντικό κοινό ερευνητικό πλαίσιο γιατί θα υπάρχει επικάλυψη και σύγχυση. Um, uh, Κάτι άλλο τώρα αναφερθήκατε και είπατε ότι δεν δώσαμε την συνέχεια στην έκθεση Καρβάλιο για τη διαδικασία της απλοποίησης. Μα ταχύτατα αναλάβαμε δράσεις ε, για να ε, ξεφορτωθούμε τους λογαριασμούς, ε, για να έχουμε καταποκοπή πόσα, για να χρησιμοποιούμε σωστό λογιστικό σύστημα για τον έλεγχο των δικαιούχων κτλ αλλά ούτως ή άλλως θα τροποποιηθούν οι κανόνες, αλλά όχι τώρα μόλις υιοθετηθεί το κοινό ερευνητικό πλαίσιο και έχουμε καταδείξει την πρόθεσή μας να απλοποιήσουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια του τωρινού ε, προγράμματος, αλλά δίκιο έχετε για την περίοδο μετά το 2013 θα πρέπει να το ε, λάβουμε και αυτό υπόψη για το κοινό πλαίσιο έρευνας και κοινοτομίας η συνεργατική έρευνα θα πρέπει να είναι το ψωμοτήρι του κοινού ερευνητικού πλαισίου στο μέλλον. Ε, καλά τα λέτε, ε, διότι χάρη σε αυτή μπορούν ε, να συναντηθούν εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων κτλ. Μετά μας είπατε για την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Ναι, προσοχή. Ε, συγγνώμη, για την προσέγγιση από, κάτω προς από πάνω προς τα κάτω πρέπει να συνδυαστεί με την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω γιατί και ε, τα δύο συστήματα έχουν τη σημασία Ε, η πολυτομεακή προσέγγιση, συμφωνώ και γι' αυτό. Αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Μιλήσατε επίση για το σημαντικό ρόλο των μικρομεσαίων. Ε, Βεβαίω, ε, ε, έχουμε στόχο 50% προ το παρόν και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα καταφέρουμε. Μιλάμε για 20.000 μικρομεσαίε επιχειρήσει που θα υποφεληθούν από ενωσιακή χρηματοδότηση. Είναι απίστευτο ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Η κυρία Καρβάλιο. Ε, είπατε θέλουμε καλύτερη διακυβέρνηση για τη χρηματοδότηση αλλά πρέπει να αναλάβουν ε, τα κράτη-μέλη το δικό τους κομμάτι. Δίκιο έχετε, δεν το έχουμε εξετάσει επαρκώς. Κυρίως ε, για τον κοινό προγραμματισμό θα πρέπει για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας να εξετάσουμε και αυτό το θέμα. Θα το μελετήσουμε λοιπόν, κυρία Μαρκής τονίζατε πόσο σημαντική είναι αυτή η μονοαπευθυντική γενιαία θηρίδα, το One Stop Shop. Ε, μα ακολούθησε τις ε, πρωτοβουλίες, τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ένωσης και προφανέστατα θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Λοιπόν, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με την Πράσινη Βίβλο τώρα την Παρασκευή που μας πέρασε. Κλείσαμε ε, το, την ηλεκτρονική μα θηρίδα. Έχουμε πάρει χιλιάδες απαντήσεις από τη διαβούλευση και τι βλέπουμε ότι ε, δεν ζητάνε μόνο τα πανεπιστήμια χρήματα για τα σχεδιάκια τους, τα προγραμματάκια τους. Έχουμε και στρατηγικά έγγραφα, λάβαμε στρατηγικά έγγραφα, όπου βλέπουμε ότι στα πλαίσια της ε, γενικότερης συζήτησης για την Ευρώπη 2020 αναπτύσσονται συνεργασίες ευρύτατες και ε, λειτουργούν πολύ καλύτερα οι διαβουλευσει και πιστεύω ότι συμφωνούν και οι πολίτε ότι είναι σημαντικό στοιχείο έρευνα και καινοτομία για την εκπλήρωση τη πολιτική 2020. Ε, τώρα ο συνδυασμός με τις έρευνας με την καινοτομία θα ενισχύσει τις γνώμες μας στην επιστημονική βάση γνώσεων και τα λοιπά. Σωστά όλα αυτά που είπατε. Στις 10 Ιουνίου στις Βρυξέλλες έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση και όλοι έχουν ε, ε, προσκαλούμε ε, όλα τα μέλη φυσικά του Κοινοβουλίου για, ε, ως συνέχεια της διαδικασίας διαβούλευσης. Περιμένουμε με ανυπομονησία την ψήφιση του σχεδίου έκθεσης της κυρίας Ματία το Σεπτέμβρη και μετά θα καταθέσουμε την αναθεωρημένη μας πρόταση για την έρευνα και την καινοτομία και στις 13 Νοεμβρίου θα πάρετε την πρότασή μας και εσείς και το Συμβούλιο. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα, οπότε περιμένουμε τη δική σας την έκθεση ε, το Σεπτέμβρη για να μπορέσουμε και εμείς ε, να συμβάλλουμε, να αρχίσουμε να συντάσσουμε το νέο σχέδιό μας ε, για να τοποθετηθείτε και εσείς ε, στη συνέχεια για το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη. Ευχαριστώ και το τελευταίο ήταν και το καλύτερο που είπατε γιατί μας παίρνετε και σοβαρά και σας ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτάκι κυρία Ματίας το πολύ γιατί έχουν σχολάσει και οι διερμηνείς. Ναι, ναι, πρόεδρε, βεβαίω. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και του διερμηνεί για το 1,5 πρόσθετο λεπτό που μας παραχώρησαν. Δεν προλαβαίνω φυσικά να απαντήσω στις ερωτήσεις και τα σχόλια που ακούσαμε. Ήθελα μόνο να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους, για τις προτάσεις τους, για τις ερωτήσεις τους. Σας ευχαριστούμε επίσης για την καλή συνεργασία Ευχαριστώ τους συναδέλφους από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θα συνεχίσουμε τη δουλειά. Είναι στενό το χρονοδιάγραμμα. Παρόλα αυτά θα τα καταφέρουμε. Μόλις τώρα το αναφέρατε. Αλλά ε, θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση. Ε, λείπει ένα πράγμα, λείπουν κάποια στοιχεία στο σχέδιο που υπέβαλα αλλά ξέρετε, όταν τριπλάσια η έκθεσή μου την ε, περιέκοψα ε, και κάποια στοιχεία σχετικά με την απλούστευση και άλλα που ανέφεραν οι συνέδελφοι ότι λείπουν από την έκθεση ήταν στο πρώτο σχέδιο. Τέλο πάντων, θα δούμε στο επόμενο. Ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. 15 εκ του προθεσμίου της Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε.